Good afternoon, colleagues. I'm going to make a prompt start because we have a uh, very tight. Um, έχουμε ένα στριμωγμένο πρόγραμμα σήμερα. Items and some votes. Και έχουμε και ψηφοφορίες. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ξεκινήσουμε χωρίς καθυστέρηση. Ανακοινώσεις του Προέδρου. δεν έχουμε κροατική, ε, μαλτέζικα και γοιδελικά. Είναι μια σημαντική ανασύνωση που θέλω να κάνω. Έγκριση δηλαδή των συστάσεων των συντονιστών της 23ης Οκτωβρίου. Σύμφωνα με το 205.2, οι πράσινοι ζήτησαν ονομαστική κλίση για την απόφαση των συντονιστών να μην οργανώσουν αποστολή στην Ουγγαρία. Το 2.4 της ημερήσιας διάταξης της συνάντησης 23 Οκτωβρίου. Η ψηφοφορία αυτή θα γίνει σήμερα στις 6 το απόγευμα. Μαζί με τις άλλες ψηφοφορίες τις οποίες θα ξεκινήσουμε. και θα εγκρίνουμε λοιπόν και αυτή την απόφαση των συντονιστών, τη σύσταση. Τώρα έχουμε την έγκριση του χρονοδιαγράμματος συνεδριάσεων για το 18. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις θεωρείται δεκτή. Έχουμε τις εφαρμοστικές και κατεξουσιοδότηση πράξεις της 26 Οκτωβρίου 2017 για το πρόγραμμα του 2018 σχετικά με τη χρηματοδότηση του προγράμματος για τα δικαιώματα, την ισότητα και την ιδιότητα του πολίτη. Πρόκειται για, την, για τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1381 του 13 σχετικά με τη δημιουργία ενός προγράμματος για την περίοδο 14-20. Η αποδοχή αυτής της εφαρμοστικής πράξης θα ανακοινωθεί σε όλα τα μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ στα πλαίσια της Επιτροπολογίας και ε, θα τεθεί προθεσμία για κατάθεση αντιρρήσεων στην γραμματεία της ΛΥΜΠΕ πριν από τις 10 Νοεμβρίου του 2017. Στις 27 Οκτωβρίου του 2017 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε μια σύσταση εξουσιοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις χώρες υψηλού κινδύνου, τις τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου που βρίσκονται στο σημείο 1 του παραρτήματος. Αναφορικά με την Οδηγία 2015-849 σχετικά με την πρόληψη της χρήσης του χρηματοοικονομικού συστήματος ε, για το πλήσιμο βρώμικου χρήματος και την χρηματοδότηση τρομοκρατικών ενεργειών. Λοιπόν, η περίοδος ελέγχου θα κρατήσει ένα μήνα και θα είναι επεκτάσιμη κατά ένα επιπλέον μήνα αν υπάρχει δυνατότητα, υπάρχει δυνατότητα κατάθεσης αντίρρησης μέχρι τις 15 Νοεμβρίου. Λοιπόν, η ηλεκτρονική ψηφοφορία θα ακολουθήσει στις 6 Παρακαλώ να έχετε όλη την κάρτα μαζί σας. Φτάνουμε λοιπόν στο σημείο 3. Το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη πρόκειται για μια ανταλλαγή απόψεων Νομίζαμε ότι θα είχαμε την Επίτροπο Γιουρόβα μαζί μας, αλλά οι συντονιστές θεώρησαν ότι πρέπει να γίνει μια τέτοια συνάντηση, αλλά δεν μπορούσε να είναι μαζί μας σήμερα και γι' αυτό θεωρούμε ότι έπρεπε να ενημερωθούμε παρόλα αυτά σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα το οποίο είναι δεσμευτικό μπροστά μας και να μπορέσουμε να θέσουμε τις ερωτήσεις προς τις ε, αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης, την Τίνα Άστολα, σχετικά με την πρώτη ετήσια ε, εξέταση της ε, λεγόμενης ασπίδας προστασίας ιδιωτικότητας. Έχουν διανεμηθεί κάποια κείμενα. Οι υπηρεσίες προστασίας των προσωπικών δεδομένων θα δημοσιεύσουν στο τέλος Δεκεμβρίου τα δικά του συμπεράσματα. Θα ζητήσουμε λοιπόν από την κυρία Αστόλα να μας ενημερώσει και μετά θα δώσω τα μέλη στους συντονιστές και αν υπάρχει χρόνος θα δώσω το λόγο και στα υπόλοιπα μέλη. Κυρία Αστόλα, έχετε το λόγο μέχρι 15 λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ, χαίρομαι όλου ιδιαίτερω που βρίσκομαι εδώ σήμερα και συζητώ ε, την ε, πρώτη ετήσια επανεξέταση ασπίδας προστασίας της ε, ιδιωτική ζωή. Όπω γνωρίζετε, το δικαστήριο κατέστησε σαφέ ότι η απόφαση καταλληλότητα δεν είναι κάτι που πρέπει να ξεχαστεί απλώ κατόπιν εγκρίσεώ τη και επομένω αυτή η υποχρέωση επανεξέτεση έχει έχει ληφθεί, έχει, η απόφαση αυτή τη επανεξέταση έχει ληφθεί στο πλαίσιο τη GDPR. Η ετήσια επανεξέταση λοιπόν τη ασπίδα προστασία τη ιδιωτικότητα είναι μία από τι βασικέ απαιτήσει του νέου αυτού πλαισίου και η παρακολούθηση είναι κάτι που τη λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη είναι αποτέλεσμα μιας πολύ περιεκτικής ε, διαδικασίας. Είναι κάτι το οποίο δεν ξεκίνησε το ε, Σεπτέμβριο στη Ουάσιγκτον. Είχαμε προετοιμαστεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα. Λάβαμε στοιχεία και από εταιρείε που συμμετείχαν σε αυτή την ασπίδα προστασίας ιδιωτικότητας και διάφορους φορείς που μας έδωσαν πολλές πληροφορίες για το πώς λειτουργεί στην πράξη και ως προς τις εταιρείε αλλά και πώς υποχρεώσεις ε, των Αμερικανικών ε, ε, αρχών ε, πράγματι γίνονται ε, σεβαστές. Έγινε λοιπόν μια πρώτη επίσκεψη στις Ηνωμένε Πολιτείε τον Ιούλιο και λάβαμε και πολλές πληροφορίες και επεξηγήσεις από τις ενδιαφερόμενες αμερικανικές αρχές. Πρέπει να πω επίσης ότι η ετήσια επισκόπηση προετοιμάστηκε και διενεργήθηκε σε πολύ μεγάλη συνεργασία με τους εκπροσώπους των αρχών προστασίας δεδομένων των κρατών μελών ε, και ε, της ομάδας εργασίας του άρθρου 29. Συναντηθήκαμε πολλές φορές πριν από την ε, συνεδρίαση της, του Σεπτεμβρίου για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την προετοιμασία μας για την ε, επίσκεψή μας στη Ουάσιγκτον ε, και φυσικά όλες αυτές, όλη αυτή η συνεργασία και τα στοιχεία που λάβαμε, ε, όλοι οι φορείς και όλες οι εταιρείε μας έστειλαν πολλά στοιχεία. Η εμπεριγνωμοσύνη των φορέων ήταν πάρα πολύ χρήσιμη για την προετοιμασία μας εν ώψη αυτής της συνάντησης, η οποία βέβαια ήταν επίσης πάρα πολύ χρήσιμη διαδικασία και ήταν κάτι το οποίο αναγνώρισε και η Αμερικανική πλευρά, η σημασία της επισκόπησης δηλαδή για τη συνέχιση της ύπαρξης του πλαισίου. Ε, φάνηκε επίσης και στο επίπεδο συμμετοχής ε, και εμπλοκής των Αμερικανικών αρχών ε, ήταν πραγματικά κάτι το άνευ προηγουμένο. Ε, ήταν ανώτατοι αξιωματούχοι παρόντες όλων των αρχών που είναι υπεύθυνε για τη διαχείριση, την εποπτεία και την επιβολή ε, και των κυβερνητικών αλλά και των πλακτικών λειτουργικών πτυχών της ασπίδας. Ε, η Επιτροπή Εμπορίου, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου, όπως επίσης ο ενεργεία διαμεσολαβητής, μέλη της, των μυστικών υπηρεσιών όπως επίσης και ε, τα μέλη του αποκαλούμενου P-Club. Ε, τα στοιχεία λοιπόν αυτά ήταν πάρα πολύ σημαντικά γιατί μας επέτρεψαν να δούμε την εφαρμογή ε, της ασπίδας. ήρθαμε πρώτα σε ε, επαφή προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι υπήρχε ανταλλαγή απόψεων πολύ καλή της ομάδας του άρθρου 29 με τους ε, εκπροσώπους των Ηνωμένων Πολιτειών. Μετά, μια πρώτη, μετά από μια πρώτη αξιολόγηση έγινε μια ενημέρωση και μετά υπήρξε μια διαδικασία ερωταποκρίσεων ε, με πολλή συζήτηση μεταξύ των δύο αντιπροσωπιών. Δεν ήταν δηλαδή απλώ μια επίσημη διαδικασία που κάποιοι φοβούνταν ότι θα μπορούσε να είναι και μπορείτε να το δείτε αυτό και από την έκθεσή μας. Επειδή ήταν η πρώτη ετήσια επανεξέταση, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποτελέσει προηγούμενο για τις μελλοντικέ επανεξετάσεις και ως προς την προετοιμασία και ως προς την ουσία της. Θα ήθελα τώρα να περάσω τώρα στα συμπεράσματα όσον αφορά τις ε, εμπορικές πτυχέ, Θεωρούμε ότι το σύστημα λειτουργεί εύρυθμα. Οι Αμερικανικές αρχές ε, έχουν δημιουργήσει τα μέσα και τους μηχανισμούς επί των οποίων είχαμε συμφωνήσει πέρσι. Καλύπτουν το σύνολο των ζητημάτων ε, από τη συμμετοχή των εταιρείων που συμμετέχουν στην ασπίδα, δηλαδή από την πιστοποίηση μέχρι την παρακολούθηση της συμμόρφωση των υποχρεώντιών τους, την επεξεργασία των καταγγελιών, όπως επίση, και, την, ε, και τη διαδικασία επιβολής. Πάνω από 2.400 εταιρείες συμμετείχαν στο σύστημα ε, και θυγατρικές ε, σημαντικών ευρωπαϊκών εταιριών. Κατά τη διάρκεια λοιπόν αυτού του χρόνου πρώτης λειτουργίας της ασπίδας, οι Ηνωμένε Πολιτείε προσπάθησαν να δημιουργήσουν τις απαραίτητες προϋπόθεσεις για την λειτουργία της ασπίδας και χαιρόμαστε βεβαίως ιδιαιτέρως ε, ότι σε σχέση με την, το παλιό πλαίσιο του ασφαλούς λιμένα τώρα γίνεται πολύ πιο αποτελεσματικός έλεγχος κατά πόσο, του κατά πόσο όντως οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από την πιστοποίηση των εταιριών γίνονται σεβαστές. Όμως πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να υπάρχει κάποια βελτίωση γι' αυτό έχουμε πολλές ε, συστάσεις συμπεριλάβει στην έκθεσή μας, ειδικότερα όσον αφορά την ε, πιο ε, προορατική και πιο τακτική παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις μετά την επιστοποίηση των εταιριών. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να πούμε ότι η νέα ε, κυβέρνηση να μπορεί να επιβεβαιώσει τις υποχρεώσεις που είχαν αναλυφθεί στο πλαίσιο της κυβέρνησης Ομπάμα Δηλαδή μιλώ για την PPD 28, ε, την Προεδρική Οδηγία Πολιτικής Υπαριθμών 28. Ε, αυτό είναι μια, ε, ένα βασικός, ένας βασικός θεμέλιος λίθος στον οποίο βασίζεται όλο αυτό το οικοδόμημα της ασπίδας προστασίας ιδιωτικότητας. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό η Προεδρική Οδηγία Πολιτικής Υπαριθμών 28 να ισχύει σε όλες τις μυστικές υπηρεσίες και την εποπτεία των επικοινωνιών αλλοδαπών βασικών μυστικών ε, ε, ε, υπηρεσιών. Κατά την ετήσια επανεξέταση, επιβεβαιώθηκε και η αξιολόγηση που έγινε κατά την περίοδο της απόφασης καταλικότητας, δηλαδή ότι παραμένουν ενισχύ κάθε πρόσβαση για λόγους εθνικής ασφαλείας από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε δεδομένα που έχουν διαβιβαστεί για εμπορικούς λόγους από την Ευρωπαϊκή Ένωση πάντοτε αποτελούσε ε, στόχο είτε μέσω εθνικών επιστολών, ε, επιστολών εθνικής ασφαλείας είτε ε, μέσω αποστολής ενός email υπό του τμήματος, υπό την έννοια ε, της υπαριθμών 702 ε, σύστασης της, του νόμου περί παρακολούθησης επικοινωνιών αλλοδαπών υπηρεσιών πληροφοριών, του νόμου ΦΙΖΑ δηλαδή. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό στο πλαίσιο της του νόμου αυτού ε, ΦΙΖΑ ε, και της, ε, του σημείου 702 είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι η περαιτέρω χρήση των δεδομένων δεν πρέπει να γίνεται αδιακρίτως και σε πολύ γενικό επίπεδο. Πρέπει να παραμείνουμε ε, πολύ προσεκτικοί και να παρακολουθούμε πολύ στενά τις εξελίξεις. Ε, η δουλειά μας δηλαδή δεν τελειώνει με τη δημοσίευση της έκθεσης αυτής και αυτό αφορά όλος ιδιαιτέρως ε, το σημείο 702 του νόμου Pfizer, του νόμου περί παρακολούθησης επικοινωνιών αλλοδαπών υπηρεσιών πληροφοριών, όπως είπα και προηγουμένως, όσον αφορά τώρα την ε, χρήση του 702 που είναι ε, η βασική, ο βασικός ε, νόμος που διέπει ε, την παρακολούθηση των επικοινωνιών αυτών. Ελπίζουμε ότι το Κογκρέσο θα, όντως θα εγκρίνει την προστασία που προβλέπεται από την οδηγία υπαριθμών 28 στο πλαίσιο της ΦΑΙΖΕ για να, μπορέσουμε να, να, μπορέσει να συνεχίσει να υπάρχει η προστασία που προβλέπεται και θα θέλαμε και εσείς να το λάβετε αυτό υπόψη υπόψη ε, στις επαφές σα με τα μέλη του Κογκρέσου. Όσον αφορά τώρα τη θέση του διαμεσολαβητή, η οποία πρέπει να ε, καλυφθεί, πρέπει να υπάρξει ένας μόνιμος διαμεσολαβητής, αυτό ήταν μία από τις βασικές ανησυχίες που προέκυψαν από την επίσκεψη της αντιπροσωπείας ΛΥΜΠΕ ε, στις Ηνωμένε Πολιτείε τον Ιούλιο. Όπως θα γνωρίζετε ενδεχομένως, ε, πολλοί πολιτικοί διορισμοί ε, έχουν καθυστερήσει στο πλαίσιο της νέας κυβέρνησης. Πάντως, Είναι μια πάρα πολύ σημαντική θέση. Η ενεργεία, η ενεργεία διαμεσολαβήτρια μπορεί να πάρει τις απαραίτητες αποφάσεις αν υπάρξει οποιοδήποτε μηχανισμός στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ενωμένων Πολιτειών που θα δρομολογηθεί. Πρέπει πάντως να ε, εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία ε, του διαμεσολαβητή ε, και αυτό μάλιστα να ελέγχεται με την εποπτεία ανεξάρτητων φορέων και να είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματα της εποπτείας αυτής και, στις και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο παρελθόν ε, η ομάδα άρθρου 29 έχουν λειτουργήσει και συνεργαστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό για να μπορέσουν να, επι, επισπεύσουν και να βελτιώσουν τη συνεργασία ε, στο πλαίσιο αυτό. Είναι όμως πάρα πολύ σημαντική η θέση του διαμεσολαβητή, γι' αυτό κάνουμε έκκληση στη κυβέρνηση των ΗΠΑ να κάνει το μόνιμο διορισμό ε, το συντομότερο δυνατόν, γιατί είναι μία από τις υποχρεώσεις, ε, μία από τις πολιτικές υποχρεώσεις ε, των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως θα είδατε, το ίδιο ισχύει και για το διορισμό των μελών του Συμβουλίου Εποπτείας της Προστασίας του Ιδιωτικού Βίου γιατί υπάρχουν κάποια μέλη που δεν έχουν διοριστεί ακόμη και ένα τέτοιο διορισμό βέβαια θα βοηθήσει την πρακτική λειτουργία τη ε, ασπίδα. Αν δεν γίνει κάτι τέτοιο ε, ή αν ε, τα θεμέλια της ασπίδας δεν παραμείνουν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βεβαίως θα αξιολογήσει εκ νέου την κατάσταση και θα ε, εξαγάγει τα απαραίτητα αποτελέσματα. Θα ήθελα επίσης να τονίσω τέλος ότι κατά τη γνώμη μα, ε, η διαδικασία αυτή επανεξέταση επανεξέτασης ήταν ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα συνεργασία εντό Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το ψήφισμα του περασμένου Απριλίου συμμετείχε. Η αντιπροσωπεία τη ΛΥΜΠΕ ε, συνεργάστηκε με ε, εταίρους ε, της ε, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Ουάσιγκτον καταφέραμε να περάσουμε πολύ σημαντικά μηνύματα. Βεβαίως όλη αυτή η διαδικασία μας βοήθησε και εμάς πολύ στην προετοιμασία της έκθεσής μας. Ήρθαμε πάρα πολύ, σε πάρα πολύ στενή συνεργασία με τις Εθνικές Αρχές Προστασίας Δεδομένων. Συμμετείχαν πολύ ενεργά στην όλη διαδικασία και βεβαίως διενεργούν και εκείνη τη δική τους αξιολόγηση. Ε, όπως είπε μάλιστα και η Επίτροπος Γιούροβα ε, πράγματι ήταν ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα του πώς μπορεί η Ευρώπη να λειτουργήσει ομαδικά. Θα ήθελα να συνεχίσει αυτή η συνεργασία, κύριε Πρόεδρε, και με πολύ χαρά θα ακούσω τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. Thank you very much, Ευχαριστώ πολύ, κυρία Στολά. Δεν είναι παροντέ όλοι οι συντονιστέ θέλουν να πάρουν αυτή πρώτο το λόγο, αλλά θα δώσω πρώτα το λόγο στου ε, συναδέλφου. Παρακαλώ περιοριστείτε στα δύο λεπτά, γιατί πρέπει να δούμε και το επόμενο σημείο στη σημερινή διάταξη στις 4 ακριβώ. Και μπορούμε να δούμε και συμπληρωματικέ ερωτήσει ε, και παρεμβάσει αν ε, υπάρξουν. Αλλά θα ήθελα να δοθούν και οι απαντήσει. Οπότε α δώσουμε το λόγο με τη σειρά Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπόνι. Ευχαριστώ για όλε τι προσπάθειε που κάνετε για την εφαρμογή τη ασπίδα προστασία ιδιωτικότητα. Είναι όντω πολύ σημαντική και η δομή των συστάσεων. Ε, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα τα πράγματα εκεί και είναι και αρκετά χρήσιμε οι συστάσει αυτέ. Θέλω να πω κάτι για αυτέ τι συστάσει ακριβώ. Καταρχά, η ευαισθητοποίηση. Η αύξηση ευαισθητοποίηση πώ μπορούμε να προστατεύσουμε του πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιο είναι το σχέδιο που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώς μπορούμε από κοινού να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση για όλα αυτά τα θέματα έτσι ώστε να γνωρίζουν πολύ περισσότερα πράγματα οι πολίτες για την προστασία της ιδιωτικότητάς τους. Δεύτερον, πώς αξιολογείται την πιθανότητα διορισμού του διαμεσολαβητού για την ασπίδα στις συστάσεις λένε ότι θα πρέπει να γίνει από τις ε, Αμερικανικές αρχές, αλλά είναι νομίζω ένα από τα βασικά σημεία για τη σωστή λειτουργία της σπίδας προστασίας ιδιωτικότητας. Πότε πιστεύετε ότι θα γίνει ο διορισμός αυτός. Και επίσης, πώς αξιολογείται αυτή την κατάσταση η οποία δεν είναι και τόσο καλή για μας ως, Ευρωπαίων, ως Ευρωπαίοι πολίτες. τι γίνεται με τις πληροφορίες που έχουμε για τις ε, αμερικανικές εταιρείες και τις πληροφορίες που δίνουν ε, για τις ε, πιστοποιήσεις, για τις αδειοδοτήσεις. Υπάρχει μια διαδικασία η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Κάποιες εταιρείες δεν έχουν μπει στον κατάλογο, οπότε μάλλον θα πρέπει να πιέσουμε τους ομολόγους μας στις ΙΠΑ και τις αμερικανικές εταιρείες, έτσι ώστε να μην υπάρξουν παρανοήσεις ή να μην υπάρξει κατάχρηση των δεδομένων των Ευρωπαίων χρηστών. Και ένα τελευταίο σχόλιο περιγράψατε πολύ, με πολύ ακρίβεια το πρόβλημα αυτής της ε, επαν... να... επανέγκρισης της, ε, ε, του, σημείου 702 και της πράξης Φάιζα. Σε ποια κατεύθυνση πιστεύετε ότι θα κινηθεί αυτό και πώς θα μπορούσε να συμπληρωθεί ή μάλλον ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Και ένα τελευταίο σημείο για αυτή την, το Εποπτικό Συμβούλιο για τις Πολιτικές Ελευθερίες και τα μέλη του που λείπουν. Όντως είναι πολύ σημαντικό. Τι μπορείτε να μας πείτε σχετικά με αυτό. Ε, ευχαριστώ για τα σχόλια που κάνατε. Ξέρω ότι κάνατε μεγάλη προσπάθεια, είναι πολλή δουλειά, αλλά πάντα είναι δύσκολο να πιέσουμε τους συναδέλφους από τις ΕΙΠΑ. Ξεκινήσαμε όμως κάπως και εξακολουθούν να παραμένουν κάποια εκρεμή ερωτήματα. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής θα απαντήσει η κυρία Σίπελ. Ευχαριστώ. Δεν μπόρεσα να ακούσω από την αρχή την παρέμβασή σας, αλλά από όσα πρόλαβα να ακούσω, θυμήθηκα ότι ε, διάβασα και μία έκθεση σχετικά και θυμήθηκα και τις συζητήσεις που κάναμε για τον ασφαλή λιμένα. Για χρόνια ακούγαμε κριτικά σχόλια, η Κομισιόν είχε υποβάλει την αξιολόγηση, την ετήσια έκθεσή τη και λέγαμε ναι υπάρχουν προβλήματα, αλλά υπάρχει πρόοδος, τα πράγματα βελτιώνονται, προχωρούν. Για χρόνια τα ακούγαμε αυτό. Και τελικά Δηλαδή, η κατάσταση ολοκληρώθηκε με μια μάλλον ατυχή απόφαση. Βλέπουμε τώρα τα ίδια προβλήματα, όπως είχαμε με τον ασφαλή να συνεχίζουν να υπάρχουν και με την ασπίδα προστασίας ιδιωτικότητας. Κυρίως όταν πρόκειται για περιπτώσεις όπου κάποιες εταιρείε κάνουν σαν να είναι μέλη της ασπίδας, αλλά δεν τη ζήτησαν ποτέ ή δεν έχουν εγκριθεί, δεν έχουν ελεγχθεί, αλλά ήδη χρησιμοποιούν τη διαδικασία πιστοποίησης στις ε, ιστοσελίδε τους. Ή όταν μιλούμε για τους τακτικούς ελέγχους. Τώρα λοιπόν βλέπουμε και όχι μόνο προβλήματα, βλέπουμε τα ίδια προβλήματα που αντιμετωπίζαμε για χρόνια με τον ασφαλή ημένα. Τι πιστεύετε λοιπόν ότι μπορούμε όντως να προχωρήσουμε στον τομέα αυτό και ποια είναι τα δικά σας σχέδια ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πείτε μας αν έχετε κάποιες ε, πιο σοβαρές, πιο απτές ενδείξεις από τις ε, Αμερικανικές αρχές για το ποιο είναι ο βαθμός στον οποίο θέλουν να συνεργαστούν μαζί μας ως προς αυτό. Το άλλο σημείο που ήδη έχει αναφερθεί έχει να κάνει με τον διαμεσολαβητή και το α, συμβούλιο της PCLOB. Έγινε ήδη αποστολή στην Ουάσιγκτον και ήδη είπαμε ότι δεν είναι σωστό να μην υπάρχουν διορισμένα όλα τα μέλη του Συμβουλίου. Έχει περάσει ένας μήνας και το πρόβλημα παραμένει. Οπότε, έχετε κάποια ένδειξη, κάποια στοιχεία από τις Αμερικανικές αρχές, ποια είναι τα βήματα που θέλουν να ακολουθήσουν για να βελτιώσουν την κατάσταση και να ολοκληρωθούν οι διορισμοί. Γιατί εγώ δεν θέλω να ξανάρθουμε εδώ σε ένα χρόνο και να συζητάμε τα ίδια πράγματα και να λέμε τα ίδια πράγματα. Ευχαριστώ. Η κυρία Ένετφελτ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Στέλλα για την παρουσίασή σα, Όπως και η κυρία Σίπολ, δεν είμαι απόλυτα σίγουρη και δεν εντυπωσιάστηκα ιδιαίτερα και παραπέμπεται στις συζητήσεις που είχαμε για τους ασφαλούς λιμένες, ασφαλείς λιμένες. Συγγνώμη. Εφαρμογή συνεπώς μιας ρύθμισης η οποία εξακολουθώ να πιστεύω δεν είναι απόλυτα προστατευμένη. Σε επίπεδο κοινοτομία έχουμε να κάνουμε με κάτι πράγματι το καινούριο. Από την άλλη ε, έχουμε τον κίνδυνο οι προτάσεις αυτές ε, να διαλυθούν στα δικαστήρια και οι ρήτρες προστασίας αυτές οι ασθενείς ε, δεν είναι εφαρμόσιμες. και η αντίστοιχη υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών δεν υπάρχει ουσιαστικά. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει διοριστεί από τον κύριο Τραμπ. Μην περιμένετε τίποτα από αυτή την πλευρά. Λέτε επίσης ότι οι προσλήψεις ε, καθυστερούν πολύ. Εδώ διορίζονται δεξιά και αριστερά παντού και στη συγκεκριμένη υπηρεσία βλέπουμε ότι υπάρχει καθυστέρηση. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Μας είπατε επίσης ότι ελπίζετε να υπάρξει ε, μια πιθανή επικύρωση της απόφασης η οποία είχε ληφθεί στο παρελθόν και ότι αυτό θα είναι αν θέλετε μια μοναδική ευκαιρία για την ενίσχυση των μέτρων προστασίας. Κοιτάξτε, έχουμε να κάνουμε εδώ με μια ρύθμιση η οποία παραπέμπει σε κάποιες διαβεβαιώσεις οι οποίες δίδονται από μια κυβέρνηση η οποία το μόνο το οποίο κάνει είναι να πιστεύει στις λεγόμενες εναλλακτικέ μορφές αλήθειας. Ποιος μπορεί να έχει εμπιστοσύνη σε αυτά. Νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος δεν γνωρίζει ότι υπάρχει μια διαδικασία κατάθεσης παραπώνων και γιατί να παραπονεθούν εφόσον δεν γνωρίζουν τι είναι αυτό το οποίο είναι σε ισχύ. Πώς θα παραπονεθείς για κάτι του οποίου την ύπαρξη δεν γνωρίζει. Συνεπώς λοιπόν νομίζω ότι η ρύθμιση αυτή δεν είναι ασφαλής και η εφαρμογή της είναι ακόμα λιγότερο ασφαλής. Εσείς λέτε ότι υπολογίζετε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υποστηρίξει την έκκληση που απευθύνεται στην Αμερικανική κυβέρνηση. Νομίζω ότι οι πολίτες περιμένουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει σεβαστό τον κοινοτικό νόμο και δυστυχώς δεν το κάνετε αυτό και μην ζητάτε από μας υποστήριξη. Να κάνετε απλά αυτό το οποίο πρέπει και οφείλετε να κάνετε για την προστασία των συμφερόντων των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εσάς κυρία Άστολα. Ευχαριστώ κυρία Άστολα για την παρέμβασή σας. Καλό είναι, νομίζω, το ότι έχουμε αυτή την συμφωνία του ασφαλούς λιμένος που εντάξει την καταφέραμε εν πάση περιπτώσει, κάνουμε την αναθεώρησή της, είναι καλό. Με ακούτε, με καταλαβαίνετε. Είναι καλό λοιπόν από αυτά τα, τις αρχικές ιδέες προσπαθούμε να βελτιώσουμε τα πράγματα που δεν λειτουργούν σωστά και να τα ε, διορθώσουμε. Ε, νομίζω λοιπόν ότι στα πλαίσια αυτής της όλης διαδικασίας προστασίας δεδομένων και της συμφωνίας που κάνουμε με την ΕΥΠΑ ε, νομίζω ότι μπορούμε να συμβάλλουμε ώστε να αναδιατυπωθούν λίγο τα πράγματα. Νομίζω ότι και σε πολιτικό επίπεδο είναι προφανές αυτό. Τώρα, αυτό που δεν είναι τόσο καλό για όλους εμάς είναι ότι δεν έχουμε μόνιμο διαμεσολαβητή. Εντάξει, για τους σκοπούς της ε, προώθησης της συμφωνίας υπάρχει ο ε, εκτελών χρέη ε, διαμεσολαβητού, αλλά εν πάση περιπτώσει προσωρινά οι λύσεις δεν είναι ποτέ καλές, πρέπει να έχουμε έναν μόνιμο διαμεσολαβητή για να μπορεί να κάνει τη δουλειά που πρέπει. Αυτό που θέλω εγώ να μάθω είναι, υπάρχει εντωμεταξύ κάποια καταγγελία έτσι ώστε να μπορεί κανείς να καταλάβει τι ακριβώς γίνεται. Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις όπου κάποιος μπορεί να παρακολουθήσει ώστε να καταλάβει ποιος είναι, ποια είναι η οδός που μπορεί να, να ακολουθήσει κανείς για να υποβάλει μια καταγγελία για να δούμε πού υπάρχουν κενά τα οποία πρέπει να γεμίσουμε. Και επίσης, ποιες είναι, ποια είναι τα βήματα που πρέπει να κάνουμε για να βελτιωθούν τα πράγματα συγκεκριμένα. Είναι κρίμα που η κυβέρνηση Τραμπ δεν φαίνεται να θέλει να πληρωθούν οι θέσεις, αλλά νομίζω ότι καλό είναι να είναι σαφές ότι η σημασία της κυκλοφορίας των δεδομένων δια μεταξύ ημών και των ΗΠΑ δεν θα μπορεί να γίνει εφόσον δεν υπάρχουν οι απαραίτητοι υπάλληλοι στις θέσεις τους για να μπορεί να γίνει αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών. Πρέπει βεβαίως τα πράγματα να γίνουν πιο γρήγορα αλλά σίγουρα πρέπει να τονίσουμε και τη σημασία της α, ε, ε, ανταλλαγής πληροφοριών και να εφαρμόσουμε αυτά που έχουμε υποσχεθεί και συμφωνήσει ότι θα, ε, θα εφαρμόσουμε. Και ξαναρωτώ λοιπόν ποιες είναι οι περιπτώσεις, αν υπάρχουν, καταγγελιών και τι βήματα έχουν γίνει για να καλυφθούν. Ευχαριστώ. Η κυρία Σαρτζεντίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολλοί συνάδελφοι είπαν αρκετά από θέλω να πω. Ο, είπαμε, είπατε κι εσείς κυρία Άστολο ότι ο διαμεσολαβητής είναι ε, προσωρινός. Ο οποίος βεβαίως η κυρία συγκεκριμένα είπε ότι δεν γνώριζε απολύτως καλά την ε, κατάσταση. Οι συνάδελφοι μίλησαν ε, για την ε, πίκλο που δεν έχει όλα τα μέλη της. Που σημαίνει ότι το θέμα είναι να υπάρχουν δυνατότητες προσφυγής για τους Ευρωπαίους πολίτες. Και αυτό προς το παρόν δεν συμβαίνει. Οπότε είναι σαν να ξαναζούμε από την αρχή τον ασφαλή λιμένα, ο οποίος βασίστηκε στην αμοιβαία εμπιστοσύνη. Και είδαμε ότι τελικώ δεν υπήρξε αμοιβαία εμπιστοσύνη, κατέρευσε ο ασφαλής λιμένας, τον αντικαταστήσαμε με την ασπίδα και το Ιρλανδικό Ανώτατο Δικαστήριο σε μία ε, υπόθεση αποφασίζει να δικαστεί η υπόθεση αυτή από το δικαστήριο στο Λουξεμβούργο. Στέλνεται λοιπόν στέλνονται λοιπόν οι ε, δικογραφίες στο Λουξεμβούργο και περιμένουμε την, απο, την απόφαση του δικαστηρίου. Οπότε πού είμαστε, Τι θα γίνει δηλαδή, κάτι παρόμοιο σε κάποια χρόνια, θα καταρρεύσει και η ασπίδα όπως ε, κατέρευσε ο λιμένας. Εν τω μεταξύ δεν έχει αλλάξει τίποτα για τους ε, Ευρωπαίους πολίτες και δεν έχει αλλάξει και τίποτα από την ε, Αμερικανική τεχνολογική βιομηχανία σε σχέση με τη διαχείριση των δεδομένων των πολιτών. Εμείς λοιπόν δεν θέλουμε οι πράσινοι καμία ε, έτσι, ε, διόρθωση του, ή με επανάληψη της κατάστασης με τον ασφαλισμένα, χωρίς να γίνουν σαφείς αλλαγές και διορθώσεις προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ. Κλείνουμε λοιπόν τον κατάλογο των ομιλητών. Να προσθέσω κι εγώ ένα ερώτημα. Μπορείτε να μας απαντήσετε τι είδους κενό είναι αυτό και πώς θα το καλύψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. είναι δύσκολο να καταλάβουμε ποια θα είναι η δυνατότητα πρόσβασης στα δεδομένα αυτά των υπηρεσιών ασφαλείας και επιβολής τάξης, νόμου και τάξης. Τι μπορείτε να μας πείτε για την πρόσβαση αυτών των υπηρεσιών στα συγκεκριμένα στοιχεία. και να μας πείτε σε ποιο βαθμό είναι καλύτερα τα πράγματα από ότι ήταν με τους, με τους ασφαλείς λιμένες και παρακαλώ σύντομα γιατί πρέπει στις 4 να τελειώσουμε. Thank you for the Some of the... Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Κάποιες είναι γενικού τύπου, κάποιες πιο συγκεκριμένες. Να ξεκινήσω από την βασική ερώτηση. Αν έχουμε μπροστά μας για μια ακόμη φορά μια διαδικασία ασφαλής λιμένες ή όχι. Κοιτάξτε, εμείς είχαμε την απόφαση για τους ασφαλείς λιμένες μπροστά μας και κάναμε και την ανάλυση των Αμερικανικών νομικών ρυθμίσεων για την πρόσβαση στα δεδομένα. Το είδαμε αυτό και στα πλαίσια του Safe Harbor. και στα πλαίσια της συζήτησης που είχε γίνει για το Safe Harbor νομίζω ότι οι απαντήσεις οι οποίες είχαν δοθεί σας κάλυπταν. Αυτή είναι μια γενική παρατήρηση βέβαια. Να περάσω τώρα στις συγκεκριμένες ερωτήσεις και να είμαι πιο συγκεκριμένη κι εγώ. Πρώτον, σχετικά με τη συνειδητοποίηση του προβλήματος. Εμείς την Άνοιξη του 18 ήδη έχουμε ξεκινήσει για τα λεγόμενα GDPR εγώ πιστεύω ότι όταν οι πολίτες συνειδητοποιήσουν ποια είναι ξεκάθαρα τα δικαιώματά τους και στην Ευρώπη, θα κατανοήσουν ότι μπορεί να τίθεται ένα θέμα και για τα δεδομένα τα οποία χρησιμοποιούνται από τις Ηνωμένε Πολιτείες. Οπότε εδώ το θέμα της ασπίδας ιδιωτικής προστασίας ε, γίνεται κάτι το πολύ πιο απτό. Υπάρχει δυνατότητα λοιπόν μέσω των GDPAs να προωθηθεί η διαδικασία αυτή συνειδητοποίησης του θέματος και υπάρχει και ένα συγκεκριμένος κατάλογος οδηγιών. Νομίζω λοιπόν ότι ο συνδυασμός των εθνικών αρχών από τη μία και των οδηγιών μας από την άλλη θα βοηθήσει τώρα για τον Ombudsman. Αυτό είναι μια απόφαση την οποία θα πρέπει να λάβει η Αμερικανική κυβέρνηση Μπορούμε να τους πιέσουμε βέβαια, το έχουμε κάνει αυτό εδώ και καιρό. Εμείς είχαμε πει ότι το θέμα αυτό είναι σημαντικό και το Κοινοβούλιο και εσείς το έχετε θέσει. Και όταν πήγαμε στις Ηνωμένε Πολιτείες το θέσαμε το θέμα ως μείζον, ως σημασίας. Πήραμε κάποιες διαβεβαιώσεις σε σχέση με τις διαδικασίες οι οποίες έχουν αποφασιστεί και ακόμα και ο προσωρινός υπεύθυνο για τα θέματα αυτά, ο προσωρινός ομπουτσμάν μπορεί να εργαστεί με βάση τα σημερινά δεδομένα και να βοηθήσει έτσι τους πολίτες να καταθέτουν τα παραπονά τους και τις αναφορές τους. Αυτό το οποίο έχει σημασία εδώ είναι η συνεργασία των επιθεωρητών σε διαφορετικά επίπεδα συλλογής πληροφοριών και τις αρχές οι οποίες τα διοικούν. Μπορεί να πει κανείς ότι στην ουσία όταν μιλάει ένας επίσημος από μία χώρα σε έναν άλλο επίσημο από μία άλλη χώρα υπάρχουν περιορισμοί. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι μπορέσαμε να κρίνουμε πόσο σοβαροί ήσαν αυτοί όταν οι γενικοί επιθεωρητές μας είπαν ποια ήταν τα δικαιώματά τους στη συλλογή πληροφοριών από τις υπηρεσίες των πληροφοριών. σχετικά τώρα με τις διαδικασίες πιστοποίησης και τις επιχειρήσεις οι οποίες ε, ε, ακόμα και αν δεν είχαν περάσει από τις διαδικασίες πιστοποίησης ε, δημοσιοποιούσαν το ότι ανήκουν στο λεγόμενο private shield. Εμείς ελέγχουμε αν υπάρχει μια διαφοροποίηση ανάμεσα από τη μία στο διαδίκτυο και από την άλλη στον κατάλογο των επίσημων, στο μητρό του επίσημο του Υπουργείου Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών. Πάντως υπάρχουν εταιρείες οι οποίες διεκδικούν το ότι ανήκουν σε αυτή τη διαδικασία, ακόμα και αν δεν έχουν περάσει από την διαδικασία πιστοποίησης. Θα πρέπει να αλλάξει η κατάσταση αυτή. Έχουμε ήδη δημιουργήσει <clears throat> μια διαδικασία θα έλεγα αρκετά σοβαρή στα πλαίσια της οποίας μπορεί να γίνεται ο έλεγχος τον οποίο αναφέρθηκα. Πάντως, αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε τώρα με το σύστημα που έχουμε στη διάθεσή μας είναι να λειτουργήσουμε προληπτικά Προς το παρόν βέβαια αντιμετωπίζουμε την πληθώρα ετοιμάτων για πιστοποίηση. Τώρα για το αν γνωρίζουμε το τι θα συμβεί από εδώ και πέρα να πω ότι δεν φαίνεται να υπαναχωρούμε, ούτε οι Ηνωμένε Πολιτείε δείχνουν κάτι τέτοιο. Εφόσον διατηρηθεί το 702 και αν οι ρήτρε προστασίας όπως τούτο το 28 θα συνεχίσουν να γίνονται σεβαστά, αυτό θα είναι κάτι το καλό και θα το ελέγξουμε. Um, Σχετικά με το P-Club. Ένα μέλος αυτή τη στιγμή είναι δραστήριο και άποψή της είναι ότι ακόμα και αν είναι τώρα το μοναδικό μέλος, όλα τα θέματα τα οποία θα πρέπει να ελεγχθούν από ομόφωνα από την, συγκεκριμέ... από την απαρτία της συγκεκριμένου PC Club δεν προχωρούν. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει διορίσει εν τω μεταξύ τον πρόεδρο της ομάδας αυτής, αλλά η διαδικασία αυτή απαιτεί την έγκριση από πλευρά της Γερουσίας. Προχωρά δηλαδή η διαδικασία, αλλά με αργούς ρυθμούς. Λοιπόν, ίδια προβλήματα που είχαμε και με το Safe Harbor. Έθεσα το θέμα κάποιων εταιριών οι οποίες υποστηρίζουν, υποκρίνονται ότι είναι μέλη της διαδικασίας Private Shield. Αλλά όπως είπα υπάρχουν αρκετοί μηχανισμοί τώρα οι οποίοι σε επίπεδο πληροφορικής μας δίνουν την δυνατότητα να ελέγξουμε αν πράγματι οι επιχειρήσεις ψευδολογούν. κάτι άλλο έχω σημειώσει εδώ, αλλά δεν καταλαβαίνω πολύ καλά τι είναι. Τώρα για το αν μπορούμε να πιστέψουμε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε θα λειτουργήσουν διαφορετικά στην περίπτωση αυτή από ό,τι είχαν λειτουργήσει στην περίπτωση του ασφαλούς λιμένος. Η απόφαση αυτή και η πρόταση αυτή βασίζεται στο safe harbor. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε δει τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο. Και ο διάλογος τον οποίο έχουμε τώρα με τους επισήμους από την άλλη πλευρά δείχνουν ότι και από δική τους πλευράς πιστεύουν ότι αν πράγματι το σύστημα δεν λειτουργήσει μπορούμε να τους ζητήσουμε να κάνουν περισσότερα και στο τέλος αν χρειαστεί να λειτουργήσουμε και με νέες προτάσεις και μέτρα. in a, in a while. However, I think that uh, the work that the US Τώρα αν αυτή η ιστορία είναι κάτι το οποίο εμεινεύεται και από τις αποφάσεις για την υπόθεση Σουέμφ, αυτό είναι κάτι στο οποίο δεν μπορώ να απαντήσω. Τώρα για το διορισμούς. Έχουν υπάρξει αρκετοί διορισμοί στις Ηνωμένε Πολιτείε. Εγώ πρόσφατα άκουσα ότι υπάρχουν 500 κενά σε διάφορα επίπεδα της διοίκησης, της κυβέρνησης, αλλά ιδιαίτερα σε σχέση με το Υπουργείο Εξωτερικών η ταχύτητα με την οποία γίνονται οι θέσεις αυτές, καλύπτονται οι θέσεις αυτές, είναι πολύ χαμηλή. Και σχετικά με το 702, εδώ το Κογκρέσο είναι αυτό το οποίο θα πάρει την τελική απόφαση. Δεν έχουν υπάρξει παράπονα μέχρι τώρα σχετικά με το πρόσωπο του Ombudsman. Εμείς συζητήσαμε να μάθουμε ποιες είναι οι διαδικασίες για να δούμε αν είναι δυνατόν να αντιμετωπίσουν τα περίπλοκα αυτά θέματα και πότε θα μπορέσουν να το κάνουν αυτό. Βλέπουμε ότι οι μηχανισμοί υπάρχουν, οι δομές υπάρχουν, δεν έχουν ακόμα επανδροθεί αλλά εδώ καλύπτεται εν μέρη το θέμα από τη δραστηριότητα των γενικών επιθεωρητών. αν έχει υπάρξει αυτό αποτέλεσμα σχετικά με το Ombudsman, με τον διορισμό του Ombudsman. Δεν μπορώ να πω διάφορα, ε, κάτι εδώ πάνω σε αυτό. Δεν νομίζω ότι οι Ηνωμένε Πολιτείες δεν αναγνωρίζουν την σημασία που έχει η υπόθεση αυτή. Είδαμε ότι έχει γίνει πολύ και σοβαρή δουλειά σχετικά με τη χορήγηση των πιστοποιητικών, με την εποπτεία, με την επιβολή των ρυθμίσεων. Αυτά όλα δείχνουν πόσο αναγνωρίζουν ότι το θέμα είναι σημαντικό. Σχετικά τώρα με το ΣΡΕΜΣ. Είναι θέμα των ρητρών προστασίας που έχουν σχέση με την κυβερνητική πρόσβαση στα δεδομένα και σχετικά τώρα με τις υπηρεσίες επιβολής τάξης. Εσείς ζητήσατε πληροφορίες από τις ε, υπηρεσίες παρόχων σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο. θα μπορούσα ενδεχομένω να πω κάτι ως προς αυτό. Είναι κάτι το οποίο αναλύσαμε διεξοδικότατα μετά τον Ιούλιο, μετά από διαμακρόν συζήτηση με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και αφορά τους περιορισμούς ε, και ειδικότερα για τις απαιτήσει ε, που υπάρχουν ε, ως προς το κόστος, για παράδειγμα, ε, που εστίασε την συγκεκριμένη έρευνα σε έναν συγκεκριμένο ύποπτο και είδαμε επίσης και τι δυνατότητες αποκατάστασης υπάρχουν. Εμείς ε, θεωρούμε ότι συνάδει με την αναλογικότητα, με την απέτηση της, προϋπόθεση της αναλογικότητας που θα έπρεπε να υπάρχει εν προκειμένου. Αυτό είναι κάτι το οποίο ε, επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους. Ε, είδαμε μία περαιτέρω βελτίωση προσφάτως η χρήση των εντολών ΓΑΚ έχουν μειωθεί. Πρόκειται για εντολές προς εταιρείες που όταν λαμβάνουν μία ε, απέτηση αποκάλυψης και πρέπει να διαβιβάσουν κάποια δεδομένα, είναι δυνατόν να ζητηθεί από τις εταιρείες αυτές να μην ενημερωθεί το ενδιαφερόμενο άτομο ε, γιατί μπορεί αυτό να αποτελεί απειλή για την ε, έρευνα όμως το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης πρόσφατα δημοσίεσε ένα έγγραφο ε, προσανατολισμού, το οποίο βέβαια συνιστά και αυτό από μόνο του βελτίωση, γιατί τώρα υπάρχει μία ε, προϋπόθεση αναθεώρησης ε, ε, αυτού του εγγράφου σε τακτική βάση και να χρησιμοποιείται βέβαια κάτι τέτοιο μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο. Αυτό προς τις διασφαλίσεις, τους περιορισμούς και τις δυνατότητες ε, ε, επανεξέτασης υπάρχει ένα επαρκές επίπεδο προστασίας κατά τη γνώμη μας, το οποίο κατά τη γνώμη μας σέβεται ε, όλα τα κριτήρια που έχουμε για να καταλήξουμε στην απόφαση περί καταλληλότητας. Κάτι ακόμη, αν μπορούσα να πω, ναι, πολύ σύντομα, για τον νόμο Φάιζα. για την παρακολούθηση των ξένων υπηρεσιών πληροφοριών. Κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μια ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας επί του θέματος αυτού. Ε, δεν συνέβαινε αυτό στο παρελθόν συχνά να έχουμε συζήτηση με τις Αμερικανικές Μυστικές Υπηρεσίες, κάτι το οποίο έγινε στο πλαίσιο ε, της ετήσιας επανεξέτασης και κατά τη διάρκεια της προσπάθειας δημιουργίας της ε, ασπίδας προστασίας και μάλιστα ήταν και ο πρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης παρών και συμμετείχε στη συζήτηση είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όσον αφορά τώρα το 702 του νόμου Φάιζα, υπάρχουν πολλές προτάσεις αυτή τη στιγμή. δεν υπάρχει μια πρόταση που να διευρύνει την δυνατότητα ε, επίβλεψης. Υπάρχει όμως ε, το US Liberty Act, ε, που συμπεριλαμβάνει εχέγγυα ε, που καλύπτουν και τους αλλοδαπούς. Αυτό νομίζω ότι είναι ε, κάτι το οποίο εισήχθη από τα μέλη του Κογκρέσου στην νομοθετική διαδικασία και είναι ένα είδος πρωτοβουλίας που θα έπρεπε να το υποστηρίξουμε και να ζητήσουμε και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να το υποστηρίξει. Έχετε μία, μία επερώτηση, κυρία Ίνετφελτ. Ναι. Εγώ δεν συμφωνώ ότι αυτό είναι χρήσιμο και ότι μας βοηθά. Θεωρώ ότι είναι γραφειοκρατικό μπλα μπλα και ότι δεν υπάρχουν εχέγγυα για τους πολίτες. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω πού βάζει το όριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πού βάζετε το όριο. Το 2016 εγκρίθηκε αυτό, δεν ε, υπάρχει όμως ακόμη διαμεσολαβητής με την κυβέρνηση Τραμπ. Ε, εσείς ήρθατε σε επαφή με πάρα πολλούς σημαντικούς ανθρώπους, αλλά δεν υπάρχει πίγκλομπ όμως, δεν υπάρχει αυτή η επιτροπή, δεν υπάρχει διαμεσολαβητής και εσείς απλώς βασίζετε σε διαβεβαιώσεις ε, από μια κυβέρνηση που δεν είναι αξιόπιστη που βάζετε το όριο και λέτε όχι δεν πάει άλλο γιατί είναι απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν είναι συμφωνία, είναι απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εσείς απογοητεύετε τους πολίτες αν τα αφήσετε αυτό να περάσει. Δεν είναι να πιέσουμε δηλαδή το θέμα λίγο τους Αμερικανούς, πρέπει να απαιτήσουμε να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Αυτό είχαμε ζητήσει. Δεν είναι αστείο κυρία Στολα, δεν είναι αστείο. Γιατί γελάτε, δεν είναι αστείο. Εντάξει, Σοφή, καταλάβαμε. Εντάξει, κυρία Στόλα, μπορείτε να απαντήσετε. Καταρχά, θα ήθελα να πω ότι υπάρχει η P-Club, αυτή η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ζωής και Ατομικών Ελευθεριών. Απλώς δεν έχει όλα τα μέλη της, ε, προβαίνουν σε εξέταση νομοθεσία, κάνουν τη δουλειά τους. Γίνεται λοιπόν αυτή η δουλειά. Με ένα μέλος μπορούν να δημοσιεύσουν τις εκθέσεις τους, οπότε υπάρχει αυτή η P-Club αυτή η Επιτροπή. Και όπως ανέφερα, έχει διοριστεί ε, πρόεδρος και αυτό είναι ένα βήμα προς την απαρτία. Όσον αφορά τώρα το διαμεσολαβητή, ακόμη και ο εκτελών χρέη έχει όλες ε, τις... Ε, μπορεί να αναλάβει πλήρως τα καθήκοντά του, δεν υπήρξαν καταγγελίες για την ώρα όταν θα υπάρξει η πρώτη καταγγελία, τότε θα δούμε κατά πόσο λειτουργεί αυτός ο θεσμός ή όχι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την επόμενη εβδομάδα θα συναντήσουμε την Επίτροπο, ίσως στις 21 Νοεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την κυρία Στόλα και την ομάδα της, αλλά και τους συναδέλφους για τις ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνάδελφοι, επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Α, ήρθε ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μπορούμε να αρχίσουμε 4 η ώρα ακριβώ δηλαδή. Thank you very much. Thank you. Get me in a flattering cough.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 Good afternoon, colleagues. We move to point four of the agenda, recent developments in Poland. Καλησπέρα. Πηγαίνουμε στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης για τις πρόσφατες εξελίξεις στην Πολωνία και τον αντίκτυπό της στο κράτος δικαίου. Είναι εδώ ο Αντιπρόεδρος Φραντς Τίμερμαντς. Καλώς ήρθατε και εσείς και η ομάδα σας. Γνωρίζετε τι έχει συμβεί Αρχίσαμε αυτή τη διαδικασία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον, Ιούριο, τον Ιανουάριο του 2016 άρχισε να παρακολουθεί την κατάσταση για το κράτος δικαίου της Πολωνίας ε, και η διαδικασία μας οδήγησε στην σημερινή ε, συνάντηση τον Αύγουστο ήρθε, έγινε ανταλλαγή απόψεων με τον Φραντ Τίμερμαντς για το θέμα αυτό ε, εδώ στην Επιτροπή μας. Κάποιοι εξημών ήσασταν παρόντες. Θα θέλαμε λοιπόν και σήμερα να ξανασυζητήσουμε το θέμα βάσει της απόφασης της διάσκεψης των Προέδρων του Οκτωβρίου που έδωσε την εντολή στην Επιτροπή να συζητήσει το θέμα αυτό εν ώψη της συζήτησης στην Ολομέλεια που θα λάβει χώρα την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Οπότε με πολύ χαρά καλωσορίζω τον πρώτο αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για να μας κάνει μια εισαγωγή ε, εν ώψη της συζήτησης αυτής στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα απλώ να πω, επειδή βλέπω κόσμο να θέλει να πάρει το λόγο, μόλις ολοκληρώσει την εισαγωγή του ο ε, Επίτροπος ε, θα ε, καταγράψω τους ομιλητές. Δύο λεπτά έκαστος πάντως. Έχουμε μία ώρα και δεκαπέντε λεπτά για ολόκληρη τη συζήτηση. Οπότε παρακαλώ θα, είστε, να είστε, θα ήθελα να είστε πάρα πολύ έτοιμοι να τηρήσετε τα δύο λεπτά. Θα είμαι πολύ αυστηρός και θα δώσω το λόγο στον ε, Επίτροπο για 10 λεπτά για να ε, ακολουθήσουμε τον τρόπο με τον οποίο κάναμε τη συζήτηση τον Αύγουστο. Να είστε παρακαλώ πειθαρχημένοι. Ε, έχετε λοιπόν ε, κύριε Τίμερμαν στο λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πολύ που μπορώ να σας ενημερώσω για το που βρισκόμαστε με την Πολωνία και τη συζήτηση για το κράτος δικαίου. Τελευταία φορά που πήγαμε ήταν 31 Αυγούστου. Τότε σα ε, ενημέρωσα για την, ε, για την τρίτη σύσταση τη Κομισιόν προ τι πολεμικέ αρχέ για το κράτο δικαίου, την οποία στείλαμε στι 26 Ιουλίου και για την έναρξη της διαδικασίας παραβάσης στι 28 Ιουλίου. Θα θυμάστε ότι οι συστάσει ε, παρουσιάζουν τι έντονε ανησυχίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματο κάτι που θα έχει πραγματικά πολύ αρνητικό αντικτυπώ στην ανεξαρτησία τη ε, δικαστική εξουσία και θα αυξήσει το συστημικό κίνδυνο στο κράτο δικαίου. Δύο ε, νομοσχέδια εστάλησαν πίσω ε, στο Κοινοβούλιο από τον πρόεδρο τη Πολωνία και θυμίζουμε βεβαίω και την κατάσταση ενός, μιας συστηματικής απειλής στο κράτο δικαίου με τι αλλαγέ που έγιναν στο δικαστικό σώμα υπονομεύοντα έτσι την ανεξαρτησία και την ομιμοποίηση του δικαστικού συστήματος λόγω της ανασύστασης εκβάθρων ε, στα πλαίσια της, ε, του διορισμού των δικαστών. Επίσης, ε, η εκτελεστική εξουσία επιμένει να αρνείται να δημοσιεύσει τις αποφάσεις των δικαστών. Ζητούμε λοιπόν από, τους, από, τις πολιτικές, από τις πολωνικές αρχές να αποκαταστήσουν την νομοποίηση του δικαστικού συστήματος ως θεματοφύλακα του πολωνικού συντάγματος. Βεβαίως, ε, είναι πραγματικά πολύ, σημαντική, ε, πολύ σημαντικές οι επιπτώσεις ε, με βάση και την πρόσφατη νόμιμική μεταρρύθμιση. Μιλούμε για την οργάνωση των τακτικών δικαστηρίων, η οποία βεβαίω βρίσκεται σε ισχύ όπω ξέρετε και στην τελευταία συζήτησή μα, επίση σα ενημέρωσα ότι δυστυχώ η πολωνική απάντηση με βάση αυτή τη αυτή της της Κομισιόν δεν προτείνει καμία αλλαγή για να καλυφθούν οι ανησυχίες τη Κομισιόν. Τι έχει γίνει λοιπόν από τότε παρά την αποστολή τεσσάρων επιστολών στις πολωνικές αρχές από τον Ιούλιο, ζητώντας να συναντηθούμε. Λυπούμε που πρέπει να σας πω ότι αυτές οι προσκλήσεις δεν έγιναν δεκτές. Κατά συνέπεια, οι ανταλλαγές μας περιορίστηκαν σε γραπτές επιστολές. Ε, Του λεκθέντος, η πρόσκληση εξακολουθεί να είναι ανοιχτή. Εξακολουθούμε να ελπίζουμε ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε προσωπικό διάλογο με τις πολωνικές αρχές και σε ό,τι αφορά τη διαδικασία υπεραβάση, οι αρχές ε, απήντησαν αρνούμενες την ε, παραβίαση ε, τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Οπότε στι 12 Σεπτεμβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να στείλει μία γνωμοδότηση ε, αιτιολογημένη προ τι πολωνικέ αρχέ. Παραμένουμε στη θέση μα ότι η πολωνική νομοθεσία είναι αντί, αντί, αντίκειται στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, διότι προβλέπει διαφορετική συνταξιωτική ηλικία για τι γυναίκε και του άντρε δικαστέ. 60 και 65 χρόνια. Κάνει διακριτική μεταχείριση με βάση το φύλλο και αυτό έχει να κάνει με το, με το άρθρο 170 της Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη ε, Οδηγία 54-2006 για την ισότητα των δύο φύλων στην, ε, στο χώρο εργασίας. Επίσης έχουμε νομικές ανησυχίες για το ότι δίνοντας στο Υπουργείο ε, Δικαιοσύνη την δυνατότητα να, να επεκτείνει την θητεία των δικαστών, δημιουργεί ένα ε, προηγούμενο και η ε, ανεξαρτησία των, δικαστη... των, δικαστηρίων συγγνώμη, θα ε, υπονομευθεί σύμφωνα με το άρθρο 19 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από με το άρθρο 47 της Χάρτας των, Ευρω... δικαιωμάτων, των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων δεν μπορεί να υπάρχει ε, ε, ε, επιρροή στους δικαστές και στην επέκταση της θητείας τους. Καθώς επίσης και το χρονοδιάγραμμα της λήψης αποφάσεων υπονομεύει την δυνατότητα απόλυσης των δικαστών. Επίσης, η ε, διακριτική ε, εξουσία για, να, για, την, ε, για την επιρροή που έχει ο, Υπουργός, ο, ο Υπουργός Δικαιοσύνης επί, επί, μεμονωμένων δικαστών όταν έχουν να κάνουν με, υποθέσεις ευρωπαϊκού δικαίου. Περιμένουμε βεβαίω να δούμε την απάντηση των πολιτικών αρχών για να δούμε τα επόμενα βήματά μας. Τώρα, ε, για την υλοτομία σε ε, ε, δασικές εκτάσεις. Βλέπουμε ότι η υλοτομία συνεχίζεται. Μετά την εντολή του δικαστηρίου της 27ης Ιουλίου για το αντίθετο. Στις 17 Οκτωβρίου έγινε μια ακρόαση ε, ε, στο δικαστήριο όπου η Κομισιόν παρουσίασε τα επιχειρήματά της για την, ε, για την επιβολή διαμέσων μέτρων στην Πολωνία. 25 Σεπτεμβρίου η Κομισιόν ενημέρωσε το, το Συμβούλιο Δικαιοσύνης για τις σχετικές δραστηριότητες και είπαμε ότι η, το, το κράτο δικαίου είναι μια κοινή ευθύνη και βεβαίω θα πρέπει από κοινού η Πολωνία και η Κομισιόν να μπουν σε διάλογο για να βρεθεί μια λύση. Την ίδια ημέρα ο πρωινό πρόεδρο Ντούντα παρουσίασε δύο νομοσχέδια στο ανώτατο δικαστήριο για, την, για το Εθνικό Συμβούλιο Δικαστών. Η Κομισιόν εξετάζει προσεκτικά τα νομοσχέδια και παρακολουθεί στενά τι ε, συνεχιζόμενε διαδικασίε και εξελίξει σχετικά με τα νομοσχέδια αυτά. Η αξιολόγηση της Κομισιόν καθοδηγείται από τις αρχές του κράτους δικαίου και τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης που πρέπει να την χάνουν σεβασμού σε οποιαδήποτε δικαστική μεταρρύθμιση. Κυρίως την ασφάλεια της θητείας των δικαστών την, αδυνα, την αδυναμία απόλυση αυτών και την προστασία τους απέναντι σε αυθαίρετες αποφάσεις των πολιτικών ομάδων και των πολιτικών ε, δυνάμων και τη εξτελεστική εξουσία. Η ανεξαρτησία αυτή δεν έχει να κάνει μόνο με την ε, ε, ανεξαρτησία τη δικαιοσύνης σε συγκεκριμένε υποθέσει, αλλά και την οργάνωση αυτής. Πρέπει να υπάρχουν εχέγγυα και εγγυήσει έτσι ώστε να διατηρηθεί η ανεξαρτησία τη δικαστική εξουσία, που είναι απαραίτητη για να υπάρξει η εμπιστοσύνη που χρειάζεται να έχουν τα δικαστήρια σε μια δημοκρατική κοινωνία. Σε αυτή λοιπόν την φάση τη αξιολόγησή τη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει ότι κάποια θέματα αυτών των νέων, αυτό, κάποια στοιχεία αυτών των νέων νομοσχεδίων πρέπει να τύχουν περισσότερη προσοχή, γιατί γύρουν σημαντικέ ανησυχίε ό,τι αφορά τι αρχέ και τα πρότυπα που σα ανέφερα. Για παράδειγμα, το νομοσχέδιο για το ανώτατο δικαστήριο ε, καταργεί την εντολή και ε, πολύ, ε, πολύ σημαντικούς, πολύ συγκεκριμένους δικαστικούς του, δικαστές συγγνώμη, του ανώτατου δικαστηρίου συμπεριλαμβανομένου και του προέδρου του χαμηλώνοντας την, το όριο ηλικίας δεξιοδότησης. Δυστυχώ όμω, ε, σε ό,τι αφορά την απόφαση για την επέκταση τη θητεία, δεν υπάρχει ούτε χρονοδιάγραμμα, ούτε κριτήρια και ούτε ε, δικαστική αναθεώρηση τη απόφαση. Επίση, σημειώνουμε το νομοσχέδιο για το Εθνικό Συμβούλιο των Δικαστών, που δίνει στα μέλη του Συμβουλίου την, ε, την, τη δυνατότητα να διορίζονται με τον ίδιο τρόπο που και καταργεί την δυνατότητα να εκλέγονται από τους συναδέλφους τους, από άλλους δηλαδή δικαστικούς θα συνεχίσουμε να ε, αξιολογούμε εις βάθος όλες αυτές τις, ε, όλα αυτά τα στοιχεία, κυρίως και με, σε σχέση με την γνωμοδότηση που θα έρθει από την Επιτροπή Βενετίας το Δεκέμβριο. Η Επιτροπή αυτή έχει ζητηθεί από, τη, από την Κοινοβουλευτική ε, Συνέλευση της, του Συμβουλίου της Ευρώπης να συντάξει δύο γνωμοδοτήσεις για, τις, για τα δύο αυτά νομοσχέδια της Πολωνίας. Οπότε τώρα επαφίεται στι πολωνικέ αρχέ να εξασφαλίσουν ότι πριν λάβουν αποφάσει για τα δύο αυτά νομοσχέδια θα λάβουν πλήρω υπόψη τι ανησυχίε που έχουν εκφραστεί στην τρίτη σύσταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώ επίση και τι ε, επερχόμενε γνωμοδοτήσει τη Επιτροπή Βενετία. Επίση, σημειώνει η Κομισιόν ότι έχουν υπάρξει και άλλε συστάσει για τα νομοσχέδια, όχι μόνο για την Πολωνία και για το ε, Συμβούλιο, Εθνικό Συμβούλιο Δικαστών, αλλά και σε ευρωπαϊκό και διεθνέ επίπεδο. Υπάρχει πρόσφατη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου των Συμβουλίων για τη Δικαστική Εξουσία και το Συμβούλιο των Ευρωπαίων Δικαστών. Επίσης αναφέρομαι στην, πρωτα, στην πρωταρχική παρατήρηση από, την ειδική, από τον ειδικό εισηγητή του ΟΗΕ, ανεξαρτήτων δικαστών και δικαστικών, ε, τον κύριο Ντιέγκο Γκαρσία Σαγιάλ, ο οποίος επίσης πιστεύει ότι η ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας απειλείται στην Πολωνία και έχει εκφράσει σημαντικέ ανησυχίε για τα δύο αυτά νομοσχέδια, για το Ανώτατο Δικαστήριο και για το Εθνικό Συμβούλιο Δικαστών. Αυτέ οι γνωμοδοτήσεις θα πρέπει να τροφοδοτήσουν τη συζήτηση στην Πολωνία για τα δύο του νομοσχέδια. Το δύο αυτά νομοσχέδια επίσης υπογραμμίζουν τη σημασία της, ανα, ε, της δημιουργίας μιας α, αναθεώρησης ανεξάρτητης και δημοκρατικής να ξαναπώ ότι οι αρχές των κρατών μελών βεβαίως μπορούν να κάνουν δικαστικές μεταρρυθμίσεις. Αλλά όταν το πράττουν πρέπει να σέβονται το κράτος δικαίου ως ένα από τους βασικούς πυλώνες ε, πάνω στους οποίους βασίζονται ε, όλες οι συμφωνίες των κρατών μελών όταν εντάχθησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξαρτάται από, αυτό, από τα κράτη-μέλη να, δομήσουν τα δικαστικά του συστήματα για το αν θέλουν να δημιουργήσουν ένα, ένα ε, συμβούλιο δικαστικών, αλλά όταν δημιουργείται ένα τέτοιο συμβούλιο για να διασφαλίζει την δικαστική εξουσία, όπως υπάρχει στο Πολωνικό Σύνταγμα, η ανεξαρτησία αυτού του Συμβουλίου θα πρέπει να την χάνει εγγύηση σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει να ε, ελπίζει σε έναν ε, ε, καλόπιστο διάλογο έτσι ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση στην Πολωνία. Και πραγματικά λυπούμε πολύ που δεν έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα να το επιτύχουμε. Για να κλείσω, να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κυρίω τα μέλη τη Επιτροπή σα για τι συνεχεί προσπάθειε που κάνετε να τηρηθεί το, το κράτο δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που υποστηρίζετε τι δραστηριότητε Τη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στην Πολωνία. Σα ευχαριστώ. Θα περάσω του συντονιστέ Μέχρι δύο λεπτά παρακαλώ. και μετά θα ζητήσω από τον Αντιπρόεδρο να δώσει μια πρώτη απάντηση και μετά θα δώσω το λόγο στα μέλη που τον έχουν ζητήσει. Λοιπόν, αν δεν μας έχετε πει ότι θέλετε το λόγο, ζητήστε τώρα το λόγο για να κλείσει ο κατάλογος. Από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα προσπαθήσω να σεβαστώ το χρόνο. Ευχαριστώ, Αντιπρόεδρε, που είστε μπροστά μας πάλι όταν συζητούμε θέματα που άπτονται τη σωστή εφαρμογή του ε, κοινοτικού νόμου. Συζητάμε την Πολωνία σήμερα εμείς όμως είδαμε να διαδηλώνουν άνθρωποι και στη Μάλτα και στη Βουκουρέστη που ζητούν την προστασία του νόμου, ισότητα μπροστά στον νόμο και καταπολέμηση της διαφθοράς. Είναι πρώτη φορά που παίρνω το λόγο σε αυτήν την Επιτροπή από την φρικτή δολοφονία της καταγγέλουσας δημοσιογράφου Γκαλίσια στην Βαλέτα που έδειξε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η δική μου χώρα. Όπως κατανοείται λοιπόν η προστασία του νόμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι το προσωπικό για μένα και για τους εκλογές μου. Το άρθρο 2 της συνθήκης λέγει ότι η Ένωση βασίζεται στην, στον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, την ισότητα, την δικαιοσύνη, το κράτος δικαίου, και τον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Είναι οι αξίες που ενώνουν οι αρχές αυτές στην Ένωση και όχι μια απλή γεωγραφική σύμπτωση. Αλλά ποτέ δεν είχαμε ζήσει τέτοιου είδου συστηματικέ απειλές. Για την Πολωνία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ζητήσει να γίνουν σεβαστές οι συνθήκες. Αλλά το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ανησυχεί για τι εξελίξει στην Πολωνία και για την έλλειψη βούλησης της πολωνικής κυβέρνησης να εμπλακεί σε επικοδομητικό διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε σοβαρές ανησυχίες με τον προτινόμενο νόμο ε, για το Εθνικό Συμβούλιο Δικαιοσύνης. Ανησυχούμε επίσης και για το ε, νομοσχέδιο για το Ανώτατο Δικαστήριο και για τις νέες προτάσεις χρηματοδότησης των ΜΚΟ, όπως επίσης και των, των ε, νέων ε, προτινόμενων ρυθμίσεων για τη χρηματοδότηση των μέσων ενημέρωσης. Σε όλους αυτούς τους τομείς υπάρχουν ελλείψεις που δεν μπορούν να αγνοηθούμε. Πρέπει λοιπόν να στείλουμε το μήνυμα ότι εμείς δεν θα είμαστε απλοί παρατηρητές ε, ενώ υπονομεύεται το κράτος δικαίου. το θέμα ε, δεν είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, να αντιπροσωπεύει μόνο ε, τα οικονομικά, αλλά αντιπροσωπεύει την ελπίδα για τους Μαλτέζους και τους Πολωνούς και δεν μπορούμε να τους εγκαταλείψουμε. Παρακαλώ μην ξεπερνάτε τα δύο λεπτά που έχετε στη διάθεσή σας. Δεν έχουμε αρκετό χρόνο. Η κυρία Ζίπελ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε γιατί το κράτος δικαίου είναι κάτι το τόσο σημαντικό. Νομίζω ότι ο ίδιος ο Επίτροπος Τίμερμανς είναι αυτός, ο οποίος εδώ και λίγους μήνες στην Ολομέλεια είπε ότι το κράτος δικαίου είναι ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να επιβιώσει η δημοκρατία και συμφώνησα με την πρόταση αυτή. Γιατί αυτό το οποίο βλέπουμε στην Πολωνία είναι πολύ σημαντικό από ένα κράτος μέλος το οποίο δεν βασίζεται, δεν σέβεται ένα, μια νομική ρύθμιση. Το θέμα του ελέγχου των δικαστηρίων δεν είναι απλά ένας επιπλέον νόμος, αλλά είναι πυλώνας για τη δημοκρατία μας. Και κάθε κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να ε, που θέλει να αλλάζει τη δικαστική εξουσία κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής της είναι κάτι το οποίο θέτει σε κίνδυνο τη δημοκρατία. Λυπάμαι επίσης και για τον χρονισμό ο οποίος επιλέγει. Η συζήτηση ξεκίνησε στις αρχές του χρόνου και φοβάμαι ότι δεν θα τερματιστούν σύντομα οι διαπραγματεύσεις. Δεν θα βρω, ε, θα έλεγα, πολλές ελπίδες για να καταλήξει η διαδικασία αυτή και αυτό με στεναχωρεί. Βλέποντας τους πολίτες της Πολωνίας θα έλεγα ότι αξίζουν περισσότερο, βλέποντας την ιστορία της χώρας, βλέποντας ε, το πόσο σκληρά πολέμησαν ε, για την δημοκρατία, πόσο σκληρά πολέμησαν για να ζήσουν ε, ελεύθεροι και σε δημοκρατικά όργανα. Και τώρα η ίδια η κυβέρνησή τους να μην τους δίδει τις απαιτούμενες εγγύησεις. Συνεπώς λοιπόν θα πρέπει όλοι μαζί από κοινού να κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε η κατάσταση αυτή να αλλάξει και να αλλάξει σε όλα τα κράτη-μέλη γιατί ίσως υπάρχουν και άλλα θέματα σε άλλες χώρες από αυτές που ακούσαμε από την Μέτσολα. Το κράτος δικαίου βασίζεται, ε, θα έλεγα, στη δημοκρατία και σιροποιεί τη δημοκρατία για πάνω από 500 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες. Ευχαριστώ. Για τους συντηρητικούς η κυρία Στίβενς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Τίμερμαν, στις αρχές Οκτωβρίου στην Ολομέλεια αναφερθήκατε στο καταλανικό θέμα και θυμάμαι αυτά τα οποία μας είχατε πει τότε. Είχατε πει ότι η αστυνομική παρέμβαση ήταν κάτι το αναλογικό σε σχέση με το πρόβλημα. Μετά βέβαια η Ισπανία ζήτησε συγγνώμη ε, για την βία αυτή που ήταν δυσανάλογη εις βάρος των πολιτών της. Οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ουσία υποστήριξε αυτό το οποίο δεν είναι δυνατό να υποστηριχθεί. Και μετά από τη σύλληψη των υπουργών της Καταλωνίας, και την, ε, το ένταλμα για την σύλληψη και απέλαση του Προέδρου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είπε τίποτα. Και ξαφνικά όταν ψηφίζεται ένας νόμος στην Πολωνία που δεν σας αρέσει, ξαφνικά την δακτυλοδεικτείτε αμέσως. Συνεπώς λοιπόν κατηγορείται και ηθικολογείται, αλλά αυτά είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά. Τι γίνεται, μήπως έχει τελειώσει το ευρωπαϊκό όραμα γιατί δεν αντιδράτε όταν το δίκαιο παραβιάζεται στην Ισπανία. Εσείς πιστεύετε ότι κάθε φορά μπορούμε με ένα μέτρο να προστατεύουμε όποιον θέλουμε και να διακόπτει φυσικά τα μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ δεν χειροκροτούν. Παρακαλώ ε, μη χειροκροτάτε και εσείς. Η κυρία Ιντβέλτ στη θέση της Γκρίσμπεκ. Ευχαριστώ, Αντιπρόεδρε, για την εισαγωγή σας. Ελπίζω και εγώ ότι κάποια στιγμή να, υπήρξε, να υπάρξει διάλογος με την πολωνική κυβέρνηση, προς το παρόν όμως κάτι τέτοιο δεν φαίνεται ότι θα συμβεί. Διαρωτώ λοιπόν ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειες για τη συνεργασία μας με τη χώρα αυτή στον τομέα της δικαιοσύνης και της αστυνομίας γιατί ε, αν θεωρήσουμε ότι η δικαστική εξουσία της Πολωνίας σήμερα δεν θεωρείται ανεξάρτητη, τι γίνεται με τα θέματα του ευρωπαϊκού εντάλματος, σαν παράδειγμα, με την κατανομή πληροφοριών και την συνεργασία ιδιωτικών εταιριών και δημοσίων αυγών, ιδιαίτερα σε θέματα δημοσίων προμηθειών οι υπόλοιπε χώρες είναι υποχρεωμένες να υποκρίνονται ότι αναγνωρίζουν τις αποφάσεις της δικαστικής εξουσίας στην Πολωνία. Συγκεντρώνουμε την προσοχή μας στην δικαστική εξουσία και αυτό δεν είναι λάθος. Από την άλλη όμως έχουμε να κάνουμε με συστηματική παραβίαση του άρθρου 2 και σε σχέση με την ελευθερία του συνέρχεστε και σε σχέση με την ελευθερία έκφρασης του πλουραλισμού των μέσων ενημέρωσης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και γι' αυτό ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο άλλωστε να λαλάβουν όλα αυτά υπόψη. Και τέλος, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι το σώμα αυτό εμένει στο να υπάρξει ένας γενικός μηχανισμός ε, σεβασμού της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτά τα οποία είπε η κυρία Μέτσολα εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ε, ήταν σωστά. Και η κυρία Στίβεν σωστά είπε ότι το θέμα δεν είναι μόνο θέμα ε, με την Πολωνία, είναι θέμα σεβασμού των ευρωπαϊκών στάνταρτ σε διάφορες χώρες. Και γι' αυτό απαιτείται ένας γενικός μηχανισμός ως προς αυτό. Και καταλήγω, Πρόεδρε, χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει κάποιες προτάσεις για ένα τέτοιο μηχανισμό εποπτείας. Πάντως εγώ ανησυχώ για την κατάσταση που επικρατεί αν βάλουμε το κομμάτι αυτό στο εσωτερικό του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Θα πρέπει να είναι κάτι το ισχυρότερο, κάτι στο οποίο θα έχει λόγο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους της ΓΟΕ η κυρία Σπινέλη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ τον Αντιπρόεδρο Τίμερμανς. Θα ήθελα να μάθω λοιπόν τι συνέχεια θέλει να δώσει ε, στην απειλή που ξεκίνησε τον Ιούλιο για παραπομπή στο άρθρο 7 αν η πολωνική κυβέρνηση συνεχίσει να αγνοεί τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα να θυμίσω ότι εν τω μεταξύ και μετά από το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, λήφθησαν μέτρα από την πολωνική κυβέρνηση όλο και πιο περιοριστικά, όλο και πιο σοβαρά και σε επίπεδο δικαστικό. Ο πρόεδρος Ντούντα άσκησε βέτο σε κάποιες από τις προτάσεις αυτές, αλλά έχουν περάσει άλλες προτάσεις οι οποίες είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές υπήρξαν διάφορα μέτρα σε σχέση με την μετανάστευση και υπήρξε υποχρεωτικός ε, εκδίωξη υποχρεωτική των μεταναστών στα σύνορα με τη Λευκορωσία. Υπήρξαν και άλλα μέτρα τα οποία εν πάση περιπτώσει περιορίζουν την ελευθερία έκφρασης, ιδιαίτερα στις συζητήσεις που γίνονται για την πολωνική ιστορία. Ε, υπήρξαν ε, μέτρα για τον έλεγχο του διαδικτύου στα πλαίσια της, τρομοκρατικής, ε, της αντιτρομοκρατικής δράσης ε, και για το εις του Ισλάμ και υπήρξαν επίσης και σοβαρά μέτρα που ελήφθησαν από την πολωνική κυβέρνηση όπως ε, η άρνηση χορήγησης του χαπιού της επόμενης μέρας, εις βάρος των γυναικών διάφορα μέτρα, εν Οπότε τι θα κάνουμε τελικά με το άρθρο 7, κύριε Αντιπρόεδρε ιδιαίτερα εφόσον το Συμβούλιο εξακολουθεί να μην παίρνει καμία προπόφαση. Προβλέπεται άλλωστε η δυνατότητα να παγώσουν κάποιες από τις πιστώσεις που προορίζονται προς την Πολωνία. Ευχαριστώ. Η Τζούντι Σαρτζεντίνη εκ μέρους των Πρασίνων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. όλα αυτά τα στοιχεία περί κράτους δικαίου, δικαίου που αναφέρθηκε, στα οποία αναφέρθηκε ο Αντιπρόεδρος, ας πούμε και το γεγονός ε, ότι τα αναπαγωγικά και δικαιώματα των ε, γυναικών τίθενται σε αμφιβόλο. Οι πρόσφυγες ε, επαναπροωθούνται στο πολωνικό λευκορωσικό σύνορο. Να μην ξεχνάμε και το πρόβλημα της χρηματοδότησης μη κυβερνητικών οργανώσεων. Όλα αυτά πρέπει να τα πούμε και πρέπει συνεχώς να επαναλάβουμε το μήνυμα, ε, το πολύ ισχυρό του ε, Επιτρόπου. Τι κριτήρια είναι αυτά που πρέπει να ε, γίνονται σεβαστά ώστε η διαδικασία, ώστε να αποφασίσουμε ότι η διαδικασία του άρθρου 2 δεν απέφερε καρπούς και τώρα πρέπει να ενεργοποιηθεί το άρθρο 7. Κάποια ίσως, ίσως να μην ε, κατάλαβα τα ε, συμπεράσματα, αλλά τα συμπεράσματα δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε η Επιτροπή της Βενετίας να καταλήξει σε έκθεση το Δεκέμβριο. Ε, πρέπει το συμπέρασμα να είναι δικό σας και να σας υποστηρίξουμε εμείς. Έχουμε ζητήσει τέσσερις φορές διάλογο. Τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε τώρα τι πρέπει να δούμε ότι θα έχει βελτιωθεί για να αποφασίσουμε ότι δοκιμάσαμε τη διαδικασία του άρθρου 2 πολλές φορές και τώρα πρέπει να περάσουμε στο επόμενο βήμα. Ευχαριστώ κυρία Σαρτζεντίνη. Η κυρία Βίνμπερκ ε, εκ μέρους του FTD δεν είναι εδώ. Η κυρία Ζήλστρα από το ΙΕΝΕΦ e ούτε εκείνη είναι παρούσα. Κύριε Πρώτε, Αντιπρόεδρε, σας δίνω το λόγο για να απαντήσετε σε αυτό το πρώτο γύρο ερωτήσεων. Κοιτάξτε, να μην ε, δίνω λάθος ε, εντύπωση. Η κυρία Στίβενς έθεσε το θέμα της Καταλωνίας που δεν είναι τμήμα της συζήτησης αυτής, ε, αλλά θέλω να απαντήσω για δύο λόγους. Πρώτον, ε, μου είπατε ότι εγώ είπα ότι οι ισπανικές ε, αρχές ε, και η απάντησή τους στο δημοψήφισμα ήταν αναλογική. Όχι, εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα στην ομιλία μου στο Κοινοβούλιο. Είπα ότι μερικές φορές η τήρηση του κράτους δικαίου μπορεί να γίνει και με κάποια χρήση αναλογικής βίας για να το πω έτσι, αλλά δεν εννοώ βέβαια ότι έχω τις πληροφορίες θα, θα, με επιτρέπ, θα μου επιτρέπουν εμένα να κάνω κάποια αξιολογική κρίση ως προς την αντίδραση των ισπανικών ε, αρχών. Φυσικά η βία δεν αποτελεί ποτέ ε, τη σωστή απάντηση και αυτό το επαναλαμβάνω συνεχώς. Ποτέ δεν θα υπάρξει λύση μέσω της βίας. Η δεύτερη παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω είναι, νόμιζα ότι μιλούσαμε για την Πολωνία σήμερα και δεν μου αρέσει αυτό το τι θα γίνει αν. Ε, κάθε φορά όταν εγώ ήμουν ε, ε, ε υπουργό εξωτερικών, κάθε φορά που υπήρχε μία επίκριση προς τη Ρωσία, ο Ρώσος υπουργό εξωτερικών μου έλεγε και τι θα γίνει αν το ένα, τι θα γίνει αν το άλλο. Λοιπόν, κοιτάξτε, ας, για κάποια θέματα που θέσατε είναι σημαντικά, καλό θα ήταν να τα συζητήσουμε, αλλά θα συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Ας συζητήσουμε αυτό που έχουμε σήμερα στην ημερήσια διάταξη, κυρία Στίβενς, Ξέρετε ότι είμαι στη διάθεσή σας. Αν θέλετε να συζητήσουμε άλλα θέματα, κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε τη δυνατότητα να τα συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή, αλλά σήμερα μιλάμε για την κατάσταση στην Πολωνία. Και δεν είναι δυνατόν να ε, δημιουργείται ε, κάποιον, να δημιουργείται αντιπερίσπασμο μιλώντας για κάτι άλλο. Ε, πιστεύω πραγματικά ότι είναι μεγάλο λάθος σε αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει να επανέλθω στο ζήτημα που αφορά την Πολωνία. Τι ακριβώς περιμένω, γιατί πολλοί ε, Βουλευτέ με ρώτησαν πότε θα ενεργοποιήσετε το άρθρο 7 ή άλλα μέσα που έχετε στη διάθεσή σας. Λοιπόν, θα είμαι απολύτω σαφέ ε, ως προς το τι αναμένουμε από τις πολωνικές αρχέ. Καταρχά. Πιστεύουμε ότι αυτά τα δύο νομοσχέδια ε, για το Ανώτατο Δικαστήριο ε, και για το Εθνικό Συμβούλιο της, του... Ε, της Δικαστικής Εξουσίας πρέπει να αναθεωρηθούν αυτά τα νομοσχέδια γιατί για την, για την ώρα όσοι έχουν αυτή τη στιγμή σημαίνει ότι το Κοινοβούλιο θα είναι υπεύθυνο κατά κάποιο τρόπο για το τι γίνεται στη δικαστική εξουσία και επίσης υπάρχει το πρόβλημα της εξαναγκαστικής συνταξιοδότησης κάποιων δικαστών. Θα ε, ήθελα να τους το πω αυτό απευθείας ε, στο, ε, σε διάλογο μαζί τους, αλλά δεν γίνεται, οπότε το λέω μέσω ημών. Επίσης, η οργάνωση των δικαστηρίων ε, να ε, συνάδει με, τα ευρωπαϊκά, με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Ξέρετε ότι τα όρια συνταξιοδότησης ε, είναι κατά παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Επίσης, η παράταση κάποιων δικαστών, κάποιο, της θητείας κάποιων δικαστών και την πάυση κάποιων άλλων όσον αφορά την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας, θα πρέπει να μην υπάρχει εξωτερική επιρροή, να μην υπάρχει ε, δυνατότητα επιλογής των δικαστών από τον Υπουργείο Δικαιοσύνη, για παράδειγμα, ε, και το θέμα επίσης της σύνθεσης του Συνταγματικού Δικαστηρίου που ανέφερα προηγουμένως. Αυτά είναι που ζητούμε. Ε, αυτά ζητούμε από τις πολωνικές αρχές και αν δεν υπάρχει ανταπόκριση για αυτά τα θέματα που δεν τα ζητήσαμε εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι κάτι το οποίο συνάδει πλήρω με ό,τι ζητούν και άλλοι διεθνεί οργανισμοί. Πάρα πολύ σαφώ. Αν δεν υπάρχει καμία υποχώρηση ω προ αυτό από πλευρά ε, από πλευράς Πολωνών, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα άλλα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μα κάποια στιγμή στο μέλλον. Θέλετε να σα πω κάτι τώρα. Ε, δεν θα πω κάτι τώρα για αυτό το θέμα ε, και δεν χρειάζεται να σας υπενθυμίσω ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να λάβει και τις δικές του αποφάσεις. Δεν χρειάζεται την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να το κάνει. Μπορείτε, αν θεωρείτε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν το χειρίζεται καλά, να αναλάβετε εσείς την ευθύνη μιας ε, δικής σας διαχείρισης κατάστασης. Μπορείτε να το κάνετε. Η κυρία Ινέτφελτ με ρώτησε ποιες είναι οι συνέπειες ε, για την αστυνομική και δικαστική συνεργασία. Λοιπόν, γενικά η δικαστική και αστυνομική συνεργασία, εν περιπτώσει δικαιοσύνη για εσωτερικά ζητήματα σε γενικές γραμμές, εξαρτώνται από την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Το γνωρίζετε πολύ καλά κυρία Ίνετφελντ αυτό. Αν η αμοιβαία εμπιστοσύνη όλο και περισσότερο αμφισβητείται λόγω της ε, αβεβαιότητας του δικαστικού συστήματος και η συνεργασία θα καταστεί πολύ δυσχερέστερη. Οπότε θα ήθελα να ζητήσω από τις πολωνικές αρχές ε, οποιαδήποτε πηγή έλλειψης εμπιστοσύνης να την απομακρύνουν. Η ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας είναι Εξαιρετική σημασία ε, Η ανεξάρτητη δικαιοσύνη, οι ανεξάρτητοι δικαστέ είναι εξαιρετική σημασία για να λειτουργήσει αυτή η συνεργασία, αλλά και η εσωτερική αγορά αν θέλουμε να λειτουργεί ε, εύρυθμα, ε, ότι δηλαδή η ενωσιακή νομοθεσία ισχύει με τον ίδιο τρόπο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόστε με τον ίδιο τρόπο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά είναι τα σχόλιά μου ως προς τις ερωτήσεις και τα σχόλια των συντονιστών. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ε, μέλη της Επιτροπής Ελίμπε τώρα. Θα λάβουν το λόγο ε, οι συνάδελφοι με τη σειρά που ζήτησαν το λόγο. Ε, panie e, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνο μια κοινότητα σε πολιτικό επίπεδο ή σε οικονομικό επίπεδο, αλλά είναι και μια κοινότητα σε επίπεδο δικαίου. Μια κοινότητα η οποία βασίζεται στις δημοκρατικές αξίες στον τομέα της κατανομής των εξουσιών και του κράτους δικαίου. Στην Πολωνία το 84% ε, υποστηρίζει των κατοίκων της χώρας ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον σεβασμό του κράτους δικαίου. Η κυβέρνηση όμως φαίνεται ότι δεν είναι σε θέση να ξεκινήσει έναν διάλογο ουσιαστικό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό σημαίνει ότι στρέφεται εναντίον του 80% του πληθυσμού, του 84% του πληθυσμού, που θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπροσωπεύει τις κοινέ μας αξίες στις οποίες θέλουν να εμείνουμε. Κλείνοντας θα αναφερθώ σε μία επιστολή ενός πολίτη 58 ετών που αυτοχειριάστηκε, προσπάθησε να το κάνει αυτό λόγω της, α, της στάσης της κυβέρνησής μας. Το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή θέτει σε κίνδυνο τα θεμέλια της χώρας και της κοινωνίας. Επιμένω λοιπόν κύριε Αντιπρόεδρε να πάρετε σύντομα μέτρα που θα οδηγήσουν σε διάλογο με την κυβέρνηση αυτή. Και ελπίζω επιτέλους η κυβέρνηση να προχωρήσει και αυτή με τη σειρά της σε ουσιαστικό διάλογο μαζί σας. Ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αν τα πράγματα συνεχίσουν όπως το επιθυμεί η κυβέρνηση, φοβάμαι ότι τα πράγματα δεν θα βελτιωθούν. Η κυβέρνηση αρνείται ουσιαστικά να υποχωρήσει στις πιέσεις και από τους ίδιους τους πολίτες της χώρας. Αναφερθήκαμε στην προσπάθεια κάποιου ο οποίος προσπάθησε να αυτοπιποληθεί λόγω της κατάστασης η οποία δημιουργείται στην Πολωνία σήμερα. Οι πολίτες είναι έτοιμοι να θυσιαστούν και αυτό δείχνει τι συμβαίνει σήμερα. Είχαμε πάρα πολύ μεγάλες διαδηλώσεις στην Πολωνία τον μήνα Ιούλιο και υπάρχουν τουλάχιστον 600 άτομα τα οποία διώκονται στην παρούσα φάση από τις δικαστικές και αστυνομικές αρχές και δεν γίνονται σεβαστά και τα προσωπικά δεδομένα αυτών που πήραν μέρος στις διαδηλώσεις. Στην Πολωνία λοιπόν στην ουσία οι περιφερειακοί εισαγγελείς διώκουν αυτούς οι οποίοι δίδουν πληροφορίες ή καταγγέλουν προς το κοινό συμφέρον. Αυτό είναι, θυμίζει τον Orwell. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας παραπέμπει πίσω στο 1984, όπου υπήρχαν πολλά παράπονα από πλευράς των δικαστών λόγω των εκαθαρίσεων στο δικαστικό σώμα. Όλα αυτά λοιπόν σημαίνουν πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι πιστεύουμε σήμερα, γιατί μεθοδολογικά σε καθημερινή βάση οι Πολωνοί που κατανοούν την δημοκρατία όπως και οι υπόλοιπη Ευρώπη χάνουν τα δικαιώματά τους, χάνουν τα δημοκρατικά τους έθιμα και συνήθεια. Και τα έθιμα αυτά είναι όπως ο αέρας τον οποίο όλοι αναπνέουμε, είναι απαραίτητα. Λοιπόν, ενθυμίστε με από τη δική σας εμπειρία οποιαδήποτε χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στην οποία η κυβέρνηση να παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως η σημερινή πολωνική κυβέρνηση. Ευχαριστώ. Θα συγκεντρώσω την προσοχή μου στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρώτον, ακούγονται συνεχώς παράπονα ότι δεν έχετε λάβει πολλές απαντήσεις από την πολωνική κυβέρνηση. Εγώ αντίθετα πιστεύω ότι η πολωνική κυβέρνηση σας απαντά σε μόνιμη βάση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει καμία εντολή να δίδει οδηγίες στα κράτη-μέλη. Προφανώς και μπορεί να έχει άποψη για κάποια θέματα, αλλά το να πούμε ότι το κράτος δικαίου απειλείται είναι κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο και όλα αυτά είναι θέματα που άπνονται του Συμβουλίου και όχι της Επιτροπής. Εσείς στην ουσία θέλετε να πάρετε τη θέση του Συμβουλίου και αυτό είναι κατά του κράτους δικαίου το οποίο χρησιμοποιείται με ύποπτο τρόπο. Δεν θέλουμε λοιπόν επιλεκτικές μορφές δικαιοσύνης. Σαν τέος υπουργό Εξωτερικών γνωρίζετε τι σημαίνει επιλεκτική δικαιοσύνη. Δείτε λοιπόν επιτέλους την πραγματικότητα στη διεθνή σκηνή. Ένα πράγμα να σας πω ότι αυτή τη στιγμή στην Γαλλία ε, τίθενται θέματα για την ελευθερία της έκφρασης. Υπάρχουν σταυροί οι οποίοι αποσύρονται και αποκρύβονται από δημόσια μνημεία και δεν διαμαρτυρήθηκε κανείς ούτε εσείς ούτε κανείς άλλος. Ε, συνεπώς λοιπόν ε, υπάρχουν επίσης και εμπόδια που τίθενται ε, στο θέμα εκλογικών διαδικασιών στην, στην Ρουμανία. Και εκεί είσαστε σιωπηλός. Για την Πολωνία μιλάτε συνέχεια, αλλά για άλλες χώρες δεν λέτε τίποτα. Λοιπόν, αύριο έχουμε τα 100 χρόνια της επανάστασης της Μπολσεβικικής. Περιμένουμε μια δήλωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για να θρηνήσουμε μαζί της τα θύματα 100 χρόνων Επανάστασης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον Αντιπρόεδρο Τίμερμανς που παίρνει σοβαρά το ρόλο του. Η Κομισιόν είναι ο θεματοφύλακας των συνθήκων και πρέπει να φροντίζει να λύνει τέτοια προβλήματα όταν προκύπτουν. Είναι υποχρέωση της Κομισιόν, δεν είναι απλώς εκτίμηση που πρέπει να κάνει. Και νομίζω ότι ο Αντιπρόεδρος το κατέστησε απόλυτα σαφές. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν είναι έτοιμη να συνδιαλλαγεί μαζί μας η πολωνική κυβέρνηση. Νομίζω ότι στις συζητήσεις συνήθως πιο εύκολα λύνονται τα πράγματα, ιδίως όταν είναι τόσο σοβαρά όσο αυτά στην Πολωνία. Κύριε Αντιπρόεδρε, το ερώτημά μου είναι το εξής. Η πολωνική κυβέρνηση έχει εκφραστεί, ε, έχει αρνηθεί ο, να κάνει διάλογο μαζί σας και τι είδους δυνατότητες υπάρχουν για να γίνει αυτός ο διάλογος. Και επίσης, αν δεν γίνει τίποτα, τι θα συμβεί. Δηλαδή αν υπάρξει μια τακτική καθυστερήσεων. Εσείς είσαστε σε ε, θέση ή διατεθειμένοι να κλείσετε το άρθρο 2 και να δώσετε σε εμά μετά τη δυνατότητα να παρέμβουμε και να κάνουμε τα απαραίτητα βήματα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βόιτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Τίμερμανς, λέτε ότι δεν μπορεί κανείς να συγκρίνει το ένα με το άλλο. Αν είσαστε θεματοφύλακας των συνθήκων, θα, να έχει, θα πρέπει να έχετε την ίδια παρέμβαση, την ίδια διαχείριση και για το ευρωπαϊκό δίκαιο. Είπατε ότι η ανεξαρτησία της ε, δικαιοσύνης βεβαίως ε, δίνει εχέγγυα για τους δικαστικούς, αλλά η Κομισιόν δεν λέει τίποτα όταν ο κύριος ε, Μάιαρ, ο δικαστής Μάιαρ στη Δρέσδη, ε, έχασε κάποια καθήκοντα για τα ΜΜΕ και επάφθη. Λέτε ότι οι κανόνες του κράτους δικαίου στην ε, Πολωνία θεωρούνται, παραβιάζονται. Και δείχνετε ότι υπάρχουν ε, λάθη, μιλάτε για την, επικριτικά για την υλοτομία λοιπά για τη συνταξιωτική ηλικία. Για την Ισπανία όμως δεν λέτε τίποτα. Ε, βγάζετε την ώρα σας απ' έξω. Ενώ και εκεί υπάρχουν διάφορες παραβιάσεις. Και στις 4 Νοεμβρίου έχει πέξει μία ε, ε, εκπομπή στο γερμανικό ραδιόφωνο που έλεγε ότι ε, ε, μπορεί όντως να υπάρξει και μία μορφή ελαφράς ε, ή περιορισμένης βίας, εν πάση περιπτώσει, για την επίλυση τέτοιου είδους διαφορών. Δεν μπορείτε να το λέτε αυτό για άλλες χώρες, αλλά και να, να κατακρίνετε μόνο την... Πολωνία και μετά όταν προκύπτουν τα ίδια προβλήματα σε άλλες χώρες να μην λέτε τίποτα. Ευχαριστώ. Να ακούσουμε την κυρία Γκόμες. Υπό το φως των ε, νέων ε, εξελίξεων για, το, για τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή, τα λεγόμενα Paradise Papers, ζητήθηκε να διορθωθεί το πρόβλημα με βάση την αλληλεγγύη και τη δικαιοσύνη κτλ. Ε, αυτό ζητάει και το κοινοβούλιο μας. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει αν το κράτος δικαίου δεν υπάρχει σε όλες τις χώρες και αυτό ακριβώς είναι που δεν λειτουργεί αυτή τη στιγμή στην Πολωνία. Εγώ είμαι από μια χώρα η οποία, στην οποία έγινε τρομερό bullying και δεν υπήρξε Κανένα που να πει ότι παραβιάζεται το κράτο δικαίου. Ένας πρώην πρωθυπουργό καταδικάστηκε για διαφθορά, για φοροαποφυγή, για ξέπλυμα μαύρου χρήματο, ακριβώ επειδή λειτουργεί το κράτο δικαίου. Το ελάχιστο λοιπόν που περιμένω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να δράσει. Και όταν η κυβέρνηση της Πολωνίας δεν θέλει καν να μπει σε διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ελάχιστο που περιμένω από την Κομισιόν είναι να δράσει και να προχωρήσει στο, στην διαδικασία του άρθρου 7. Okay, under... Λοιπόν, αν έχουμε ε, χρόνο, ε, στο πλαίσιο του κανόνα 206, θα μπορούμε να ακούσουμε και κάποια μη μέλη της ΛΥΜΠΕ. Να ακούσουμε πρώτα την κυρία Φισνεύσκα Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με λύπη μου παρατηρώ ότι για μια ακόμη φορά η Επιτροπή μας ασχολείται με τα θέματα της απειλούμενης υποτίθεται δημοκρατίας στην Πολωνία. Κοιτάξτε, θα πρέπει να καταλάβει η αντιπολίτευση στην Πολωνία ότι έχασε τις προηγούμενες εκλογές. Πάρα πολύ απλά. Και τελικά βλέπουμε ότι η πολωνική κυβέρνηση προσπαθεί να δημιουργήσει μια ψευδή εικόνα μιας Πολωνίας η οποία έχει εξαγερθεί. Ελάτε στην Πολωνία να δείτε πώς γίνεται σεβαστός ο νόμος στην χώρα μου. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή έχει την πλειοψηφία της ε, Πολωνικής Βουλής. Να σας διαβεβαιώσω λοιπόν κύριε Τίμερμανς ότι εμείς εφαρμόζουμε απλά τις εκλογικές μας υποστέσεις. Στην Πολωνία οι Πολωνοί αποφασίζουν. Αυτή είναι η δημοκρατία, ότι δηλαδή η πλειοψηφία έχει το δικαίωμα να εφαρμόσει το πρόγραμμα πάνω στο οποίο ε, ψήφισε. Εσείς έχετε φτάσει σε απίθανα σημεία. Ισχυρίζεστε ότι υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών στους δικαστές στην Πολωνία. Να σας πω ότι κάτι τέτοιο ισχύει και σε άλλες οκτώ χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε το θέμα αυτό ε, δεν μπορείτε να το αγνοείτε, είναι λίγο παράλογες οι κατηγορίες τις οποίες μας απευθύνεται και μάλιστα και σε κάποιες δηλώσεις κομμουνιστών και σοσιαλιστών αναφερθήκαν κάποιοι συνάδελφοι από τον χώρο αυτό στα αναπορεγωγικά δικαιώματα. Κοιτάξτε, τα αναπαραγωγικά δικαιώματα ε, είναι κάτι το οποίο ανήκει στο ζωικό βασίλειο. Θα πρέπει να κάνετε τη διάκριση ανάμεσα στην απλή αναπαραγωγή από την άλλη και την δυνατότητα επιλογής τεκνοποιίας. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Πρέπει λοιπόν να σέβεστε τις δημοκρατικές εκλογές που έγιναν στην ε, Πολωνία. Και να πω εδώ στους κομμουνιστές ότι στην Πολωνία η κομμουνιστική προπαγάνδα είναι πάρα πολύ απλά απαγορευμένη και αποκομμουνιστοποιούμε τα ονόματα των δρόμων. Κοιτάξτε, σύμφωνα με το 264 Make sure um, Κοιτάξτε, είναι στη διακριτική μου ευχαίρεια να δίνω το λόγο σε μη μέλη της Επιτροπής μας. Κοιτάξτε, θα μιλήσετε εσείς τελευταία. Θα δώσω τον λόγο στην κυρία Χολμάιερ ένα μέλος, ε, μη μέλος, ένα μέλος του Κοινοβουλίου που δεν ανήκει στην ε, Λίμπε όμως πρώτα. Ο κύριος Κούσμιτς. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αντιπρόεδρε, το κράτος δικαίου στην Πολωνία είναι μια χαρά σας χαιρετά. Η δημοκρατία ανθίζει στη χώρα μου. Αλλά για μια ακόμη φορά αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιμετωπίζει την ε, κατάσταση με απαράδεκτο τρόπο. Μιλάτε για το συνταγματικό δικαστήριο της χώρας μου. Εγώ κοίταξα τις περιπτώσεις τις οποίες εξέτασε το συνταγματικό δικαστήριο μέχρι το τέλος του μηνός Σεπτεμβρίου. 400 περιπτώσεις. Πάνω σε 400 περιπτώσεις ε, ελήφθησαν αποφάσεις. Ε, δουλεύει κανονικά το δικαστήριο, οι καθυστερήσεις ε, έχουν περιοριστεί επίσης και τώρα τα πάνε τα πράγματα καλύτερα γιατί η προηγούμενη κυβέρνηση ασχολιόταν με την πολιτική και όχι με τον νόμο και τη δικαιοσύνη. Ο νόμος λοιπόν ο νέος ισχύει ε, για τα 400 δικαστήρια εδώ και τρεις μήνες και αυτοί οι οποίοι ήταν επικεφαλής των δικαστηρίων που αντικαταστάθηκαν είναι γύρω στους 10 και ότι αυτό το οποίο λέγουν οι σοσιαλιστές ότι αντικαθιστούνται όλοι οι υπεύθυνοι των δικαστηρίων είναι εντελώς ψευδές. Τώρα για την συνταξιοδότηση, την ημερομηνία συνταξιοδότησης και τη μείωση των, του ορίου συνταξιοδότησης ε, είναι κάτι το οποίο δεν θα αφορούσε αποκλειστικά στους δικαστές, γιατί οι δικαστές θα έπρεπε να δουλεύουν, αν δεν κάναμε τις απαιτούμενες αλλαγές, ε, πολύ περισσότερο από όλους τους υπόλοιπους εργαζομένους. Είναι απαράδεκτο να θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βάλει η Πολωνία να δουλεύουν οι δικαστές της πιο πολύ από ό,τι στις άλλες χώρες. Τώρα για το ανώτατο δικαστήριο. Δεν μπορούμε να το συζητήσουμε το θέμα στην παρούσα φάση γιατί πρόκειται για κάτι το οποίο εξελίσσεται συνεχώς. Λέτε να μην συζητάμε άλλα θέματα. Στην Γαλλία όμως υπάρχουν ε, διατάγματα που περιορίζουν τα δικαιώματα των εργαζομένων. Σιωπή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ισπανία στην ουσία διαλύεται πλέον η Επιτροπή Σιωπή. Λοιπόν, αν συνεχίσετε με τον τρόπο αυτό, μόνοι σας από τα μέσα θα διαλύσετε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεχάσαμε δύο συναδέλφους που ήθελαν να πάρουν το λόγο και μας το είχαν πει εντός του χρόνου που είχα προβλέψει γι' αυτό. Η κυρία Σπινέλη για ένα διαδικαστικό. Μπάρμπαρα, πάρα πολύ σύντομα παρακαλώ. Πάρα πολύ σύντομα. Θα ήθελα απλώς να επενθυμίσω στον Πολωνό συνάδελφο, καταρχάς εγώ δεν είμαι κομμουνίστρια. Ε, δεύτερον, το αποτέλεσμα μίας ε, εκλογικής αναμέτρησης ε, η πλειοψηφία δεν είναι συνώνυμο του κράτους δικαίου. Η πλειοψηφική κυβέρνηση ε, υπόκειται στο κράτος δικαίου. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Χολμάιερ. Καταρχάς να πω ότι πρέπει οι κυβερνήσεις να τηρούν το κράτος δικαίου ανεξάρτητα από το αν έχουν πλειοψηφία. Η πλειοψηφία δεν τους δίνει λόγο να είναι κατά του κράτους δικαίου. Υπάρχουν βάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τους έχουμε ψηφίσει και το κράτος δικαίου είναι μία από τις βασικές αρχές η οποία ισχύει καθολικά. Οπότε πρέπει να έχουμε πιο γρήγορο, πιο αποτελεσματικό μηχανισμό για να λύνουμε τέτοια προβλήματα. Ε, και βεβαίω και για την Ισπανία, ανεξάρτητα αν θέλουμε να προχωρήσουμε έτσι ή όχι, εκεί το πρόβλημα δεν είναι η ανεξαρτησία της, δικαστική, της δικαστικής εξουσίας. Εκεί η δικαστική εξουσία ε, κινείται με βάση το Σύνταγμα, ανεξάρτητα από το αν το θέλει ή όχι η κυβέρνηση. Οπότε πρέπει τα δύο πράγματα να τα ξεκαθαρίζουμε. Ε, ήθελα να θέσω ένα ερώτημα στον κύριο Τίμερμανς. Τα κράτη-μέλη λόγω και των αυξανόμενων ε, προβλημάτων που υπάρχουν σε ό,τι αφορά το κράτος δικαίου, είναι έτοιμα να συμφωνήσουν με έναν τέτοιο μηχανισμό όπως ε, ε, ζητά το Κοινοβούλιο ή όπως έχει προτείνει η Σόφη στην έκθεση πρωτοβουλίας της η οποία συμφωνήθηκε, ψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία για έναν πιο ακριβή, πιο γρήγορο και πιο ικανό να αντιδρά μηχανισμό γιατί πραγματικά έχουμε διάφορα προβλήματα. Υπάρχει, ο κανονισμό, υπάρχει το άρθρο 7, ε, υπάρχουν οι δυνατότητες ε, ε, διαλόγου, αλλά καμιά φορά αυτές οι, επιλογές που έχουμε δεν είναι παρκείς, οπότε θέλω να δω αν μπορούν τα κρατημέλη να συμφωνήσουν σε κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Χόνσταϊν, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. πραγματικά θλίβομαι που κάποιοι προσπαθούν να μετα τρέψουν τη συζήτηση αυτή σε προώθηση της δικής τους, ε, του δικού τους πολιτικού προγράμματος. Ε, εμείς εδώ δεν είμαστε για να προσπαθήσουμε να βλάψουμε τους άλλους, αλλά για να συζητήσουμε σημαντικά πράγματα. Και το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ δραματικό. Μία κυβέρνηση που έχει πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο, παραβιάζει τον νόμο, είναι μία δραματική κατάσταση, είναι κάτι το άνευ προηγουμένου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν χρειάζεται να επαναλάβω νομίζω ότι η δημοκρατία α, είναι ο σεβασμός του νόμου αλλά ε, και της ε, ε, αντιπολίτευσης που έχασε τις εκλογές. Πρέπει να σέβεται η κυβέρνηση αυτή όλους όσους μπορούν να διαφωνούν μαζί σου. Πάρα πολλά ζητήματα βρίσκονται ενώπιον της δικαιοσύνης στην Πολωνία σήμερα που που πραγματικά φοβούμε ότι το δικαστήριο της Ένωσης ε, θα έχει πάρα πολλή δουλειά ε, σύντομα γιατί πάρα πολλοί κόσμος θα ζητήσει να δικαιωθεί στο δικαστήριο της Ένωσης. Και ολοκληρώνοντας θα ήθελα να πω ότι πιστεύω πραγματικά ότι οι δημοκράτες όλων των χωρών, αν συνεργαστούν, ε, θα επικρατήσει η δημοκρατία σε όλη την Ευρώπη. Όσοι λοιπόν ζουν σε δημοκρατική ε, χώρα, να συνεργαστούν, να συνεργαστούμε με τους ε, μη κυβερνητικού οργανισμούς, με τους πολίτες, με τα πολιτικά κόμματα και με όλους όσους ενδιαφέρονται για τις κοινέ μας ευρωπαϊκές αξίες. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι άνθρωποι στην Πολωνία, σας διαβεβαιώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος, συνάδελφοι ευχαριστώ πολύ. Έχετε το λόγο κύριε Τίμερμαν. ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ε, ε, σχόλιά σας. Θα προσπαθήσω να τα τιμήσω με την απάντησή μου. Ε, Νομίζω τώρα το κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να χρησιμοποιήσει το πλαίσιο κράτους δικαίου, νομίζω ότι δεν είναι αυτό το θέμα, αλλά, τέτοιο θέμα, αλλά εφόσον ε, τίθεται, πρέπει να σας πω ότι ναι, ε, το πλαίσιο του κράτους ε, δικαίου είναι μια ευθύνη που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η δυνάμη του άρθρου 7, ε, μπορεί να ζητήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενεργοποιήσει τους προληπτικούς και κυρωτικούς ε, μηχανισμούς του άρθρου 7, ε, μεταξύ των οποίων βέβαια είναι και το κράτος δικαίου του άρθρου 2, δηλαδή πως είναι δυνατόν να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε παραβίαση από πλευράς κράτους μέλους του κράτους δικαίου και παραπέμπεται στο άρθρο 7. Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει ζήτημα αρμοδιότητας. Ε, δεν μπορώ να καταλάβω πώς αυτό το θέμα ανακύπτει συνεχώς. Έχετε αρχίσει να αμφισβητείτε τα κίνητρα των ατόμων που το αναφέρουν συνεχώ. Αλλά συμφωνώ με την κυρία Χολμάιερ και την ε, κυρία Ίνετβελτ ότι το σύστημα όσο έχει αυτή τη στιγμή έχει κάποια σημαντικά κενά γιατί δεν μας επιτρέπει αρκετό περιθώριο για να υπάρχει συζήτηση ε, με ε, ακόμη και εντό του Συμβουλίου. Ξέρω ότι το Κοινοβούλιο έχει πάρα πολύ σημαντικέ και ε, αποκρισταλωμένε απόψεις προ το θέμα και έχω πει πολλέ φορέ ότι είναι πάρα πολύ ε, σαφέ ότι πρέπει να συμπεριληφθεί το Κοινοβούλιο σε, σε αυτό το διάλογο και το λέω αυτό προ την κυρία Ινέτβελτ και στο Συμβούλιο υπάρχει αυξανόμενη υποστήριξη για την ιδέα την οποία προωθεί σε μεγάλο βαθμό η βελγική κυβέρνηση να υπάρχει μια ευρύτερη επισκόπηση, ας πούμε, ομοτήμων ε, για τα ζητήματα κράτους δικαίου, γιατί υπάρχει πάντοτε έτσι μια δυσαρέσκεια, μια μηχανία όταν κάτι ε, συμβαίνει σε ένα άλλο κράτος μέλος, να υπάρχει ένα άλλο κράτος μέλος που να πρέπει να το θέσει. Να υπάρχει λοιπόν μια ευρεία επισκόπηση είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή έχει περισσότερη υποστήριξη αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο από τότε που εγώ ήμουν υπουργό Εξωτερικών και το είχα προτείνει στο Συμβούλιο. Μπορούμε λοιπόν να προχωρήσουμε και στο πλαίσιο του Συμβουλίου γιατί συμφωνώ. Συμφωνώ ε, με την ανάλυση των δύο ε, κυριών που προανέφερα. Θα ήθελα να πω γιατί εστιάζεστε πάρα πολύ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να θέσαμε το θέμα του κράτους δικαίου στο Συμβούλιο, ε, υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη υποστήριξη των κρατών μελών ε, υπέρ της ε, θέσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δηλαδή η ιδέα ότι υπάρχει ένας τρελός ας πούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που επιτίθεται στην Πολωνία δεν, είναι, δεν ισχύει. Τα περισσότερα κράτη-μέλη τα θέτουν τα ζητήματα αυτά με ανησυχία. Δεν θέλουν να την τιμωρήσουν. Θέλουν απλώς να φύγει από αυτήν την ε, οδό, την επικίνδυνη, ε, να, τη να την ε, ε, οδηγήσουν εκεί που θα έπρεπε να είναι η Πολωνία, στο κέντρο της Ευρώπης. Γιατί ο κόσμος καταλαβαίνει τη σημασία του κράτους δικαίου για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της εσωτερικής αγοράς, της δικαιοσύνης εσωτερικών υποθέσεων και όλων των υπολείπων τομέων ε, που άπτονται αυτού και ειδικότερα βέβαια η προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών μας. Πρώτο και κύριο, οι Πολωνοί πολίτες είναι Ευρωπαίοι πολίτες και αξίζουν την ίδια, τα ίδια, ε, την ίδια προστασία ε, με τους υπόλοιπους πολίτες της Ένωσης. Αυτό είναι κάτι το οποίο ε, είναι ζωντανό στο Συμβούλιο. Μην θεωρείτε ότι εγώ ας πούμε έχω παραρχίσει καμία εκστρατεία κατά της, ε, της Πολωνίας. Υπάρχουν άνθρωποι και εγώ βεβαίως που με κάθε μου ιδιότητα πάρα πολύ πολέμησα για τη θέση της Πολωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε λοιπόν οποιαδήποτε επίκριση είναι κάτι την οποία συμμερίζονται σε μεγάλο βαθμό πολλά κρατημέλη. Μην απατάστε και δεν θέλουν να βάλουν στη γωνία την Πολωνία και να τη στριμώξουν, αλλά ενδιαφέρονται πραγματικά για την Πολωνία και θέλουν να επανέλθει, να επανέλθει στο δρόμο του κράτους δικαίου που έχει, έχει ως αποτέλεσμα πολλά καλά πράγματα για την Πολωνία τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι το πρώτο μου σχόλιο. Δεύτερον, το θέμα της ηλικίας συνταξιοδότησης για το γενικό θέμα της ε, η εξία συνταξιοδότησης, ε, η ίση μεταχείριση ε, είναι ένας κανόνας που υπάρχει από το 1979 σταδιακή ισότιμη μεταχείριση ανδρών και γυναικών σε ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ των οποίων και οι ηλικίε ταξιδότησης. Ένα κράτος ε, μέλος δεν χρειάζεται να το κάνει αμέσως αυτό, να ορίσει μια ε, ηλικία συνταξιοδότησης ίδια σε όλα τα κράτη, αλλά πρέπει να κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Τα κράτη-μέλη που έχουν διαφορετικά διαφορετικά, ε, διαφορετικά όρια συνταξιοδότησης για άνδρες και γυναίκες πρέπει να λάβουν βήματα προς την κατεύθυνση αυτή. Το να επανεισάγονται διακρίσεις όπως γίνεται με το νομοσχέδιο το πολωνικό περί συνταξιοδότησης δεν είναι συμβατό ούτε με το γράμμα ούτε με το πνεύμα της νομοθεσίας της Ένωσης ε, και Υπάρχει περίπτωση να αυξηθεί και η φτώχεια των γυναικών αν έχουν χαμηλότερη ηλικία συνταξιοδότηση. Αυτό είναι κάτι που έχει αναφερθεί πολλέ φορέ και στι ειδικέ αναχώρασει τάσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση προ την ε, ε, Πολωνία. Ε, η μείωση τη ηλικία συνταξιοδότηση δημιουργεί και άλλα προβλήματα, όπω για παράδειγμα την οικονομική βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματο πραγματικά έχουμε μία πραγματική ευθύνη να κάνουμε κάτι «40% είναι το χάσμα μεταξύ συνταξιοδότησης ε, ανδρών και γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με το να δημιουργούμε διαφορετικά όρια συνταξιοδότησης ε, ε, επιδεινώνουμε το πρόβλημα». Προφανώς οι γυναίκες ε, πρέπει και εκείνες να έχουν μία ευκαιρία ε, στην οικονομική επιτυχία, δεν πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους άντρες, να κάνουν ε, τις δικές τους επιλογές και να μην τους επιβάλλονται οι επιλογές αυτές πολιτικά. Νομίζω ότι αυτό είναι αναπόσπαστο τμήμα της ενωσιακής νομοθεσίας και των κοινών μας αξιών. Και κάτι ακόμη, ένα ακόμη ζήτημα το οποίο πρέπει να τονίσω γιατί αυτό ανακύπτει πολύ συχνά. Το να λέμε ότι επειδή κερδίσαμε τις εκλογές, αυτό είναι αποτέλεσμα της δημοκρατίας και μπορούμε να αποφασίζουμε τι θα πει κράτος δικαίου. Ή τι σημαίνει, τι, ποια είναι ακριβώς ε, η, έννοια του κράτους δικαίου. Δεν υπάρχει καμία νίκη σε εκλογές που σου δίνει τη δυνατότητα να παραβιάζεις ή να αγνοείς την νομοθεσία και το Σύνταγμα. Και όπως είπα και προηγουμένω, ε, κάποια στοιχεία, όπω για παράδειγμα τα θέματα του συνταγματικού δικαστηρίου, κάποιου από τους δικαστές που διορίστηκαν, διορίστηκαν κατά παράβαση ε, του, συντα... του, ε, του συντάγματος του πολωνικού δεν... και και κάποιοι που έπρεπε να είχαν διοριστεί τελικά δεν έλαβαν ε, θέση στο συνταγματικό ε, δικαστήριο. Ε, υπάρχουν πράγματα τα οποία αναφέρονται στο σύνταγμα της χώρας και δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε το επιχείρημα ότι κερδίσατε τις εκλογές για να μπορέσετε να παραβιάσετε το σύνταγμα και να ορίζετε τι θα πει κράτος δικαίου. Μπορείτε να αλλάξετε το σύνταγμα. Αυτό αποτελεί δημοκρατικό σας δικαίωμα. Η δημοκρατία, αν έχετε την πλειοψηφία σας, δίνετε δυνατότητα να αλλάξετε το σύνταγμα, αλλά να αλλάξετε το σύνταγμα δεν μπορείτε να το κάνετε στο βαθμό που αυτό παραβιάζει ε, τις αρχές ε, ε, των διεθνών οργανισμών στους οποίους έχετε προσχωρήσει, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν μπορείτε να το κάνετε επειδή έχετε τη δημοκρατική ψήφο του λαού. Αν λοιπόν ορίζεται οτιδήποτε ε, από ευρωπαϊκή ιστορία, ξέρουμε ότι το επιχείρημα της δημοκρατίας στο παρελθόν μας έχει χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση των ε, ε, δικαιωμάτων των πολιτών και την ε, ε, παραβίαση ε, του κράτους δικαίου. Δημοκρατία, σεβασμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σεβασμός κράτους δικαίου, αυτά αποτελούν τη δημοκρατία. Το ένα δεν μπορεί να χρησιμοποιείται εναντίον του άλλου αν δεν θέλουμε να ξανακάνουμε τα σφάλματα που έχουν κάνει οι Ευρωπαίοι στο παρελθόν. Και ξέρετε πολύ καλά με την πολωνική ιστορία ότι οι κομμουνιστές χρησιμοποίησαν το κράτος δικαίου κατά της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, όταν τους Ήθεστε κάτι που το έκανα εγώ, γιατί αγνοούσαν το κράτο δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα έδειχναν το, έδειχναν το σύνταγμά του και έλεγαν Μα αυτό το γράφει το σύνταγμά μα. Αν δεν θέλετε λοιπόν να χρησιμοποιεί ο κόσμο το κράτο δικαίου κατά τη δημοκρατία, τότε μην κάνετε και το αντίστροφο. Πρέπει αυτοί οι τρει πυλώνε τη ελεύθερη ευρωπαϊκή μα κοινωνία ε, πρέπει να του σεβόμαστε αν δεν θέλουμε να ξαναγίνουν τα σφάλματα του παρελθόντο. Σα εκλυπαρώ λοιπόν, σταματήστε να χρησιμοποιείτε αυτό το επιχείρημα σήμα ότι αυτό που κάνουμε είναι απλώς η μετάφραση μιας ε, δημοκρατικής ψήφου. Δεν υπάρχει καμία, ε, κανένα κόμμα ε, στην Πολωνία που να έλεγε κατά την προεκλογική εκστρατεία ότι θα έκανε μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος ή του συνταγματικού δικαστηρίου. Οπότε το να μου λέτε ότι έτσι ανταπεξέρχεστε στις υποσχέσεις προεκλογικές δεν ισχύει για όλους όσους τώρα επέκριναν τη θέση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κοιτάξτε, αυτό δεν έχει, να κάνει, δεν έχει καθόλου να κάνει με τις, ε, με τις προτάσεις που κάναμε. Ε, μιλήσατε για τις αρμοδιότητες, για το επιχείρημα της ε, δημοκρατίας, για το θέμα του, του ηλικιακού ορίου συνταξιοδότησης. Το να χρησιμοποιείτε όμως άλλα ε, θέματα ε, τα οποία χρήζουν συζήτηση. Να συζητήσουμε για τη Μάλτα, για την Καταλωνία, για ό,τι θέλετε. Εμείς δεν κάνουμε διάκριση. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Έχουμε αχρωματοψία σε αυτά τα πολιτικά ζητήματα και το έκανα και στην Ολομέλη και θα το κάνω κάθε φορά που θα χρειαστεί. Όμως, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Α μην αρχίσουμε τώρα να κάνουμε αντιπερισπασμού και να λέμε τι θα γίνει με το ένα, τι θα γίνει με το άλλο, όταν έχουμε να συζητήσουμε ένα σοβαρό θέμα που θα γίνει με το κράτο δικαίου στην Πολωνία. Δεν είναι ισχυρότερα τα επιχειρήματά σα αν χρειάζεται για να ε, μεταφέρετε την προσοχή κάπου αλλού, να χρησιμοποιείτε άλλα σοβαρά ζητήματα στο επιχείρημά σα που πρέπει να συζητηθούν. Πολλέ φορές ε, μιλήσατε για πολλά ζητήματα τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε μια πολιτική συζήτηση στην Πολωνία, για παράδειγμα αν υπάρχει πράγματι ένα νομοσχέδιο για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που θα παρουσιαστεί στο Κοινοβούλιο. Να το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή αυτό, αλλά σήμερα έχουμε να συζητήσουμε το θέμα αυτό του ε, Συνταγματικού Δικαστηρίου και των τεσσάρων ε, ε, νόμων που βρίσκονται στη διαδικασία έγκρισης στο ΣΕΙΜ, στο Πολωνικό Κοινοβούλιο. Και πρέπει να σας πω μία ακόμη φορά ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η νόμοι αυτοί είναι μία απειλή, είναι μία συστημική απειλή για το κράτος δικαίου στην Πολωνία. Το τονίζω αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δεν είναι μόνη της ε, όταν το πιστεύει αυτό. Ε, πολλοί εκπρόσωποι ε, της δικαστικής εξουσίας συμφωνούν και εκπρόσωποι της Επιτροπής του ΟΗΕ. Έχουμε μάθει πολλά πράγματα από την Επιτροπή της Βενετίας στο παρελθόν. Θα ακούσουμε και τη δική τους έκθεση σύντομα. Η πολωνική κυβέρνηση δεν μπορεί να τα γνωρίζει όλα αυτά και λένε, να λέει ότι Υπάρχει ένας τύπος εκεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχει πρόβλημα με μας και θέλει να ε, ε, μας επιτεθεί. Είναι προφανώς ότι η πλειοψηφία της κυβέρνησης ε, ε ε, γνωρίζει ότι υπάρχουν πολλές ε, ανησυχίες σε πολλά κράτη-μέλη για το θέμα αυτό. Η Γαλλία, για παράδειγμα, το έχει αναφέρει πολλές φορές. Άλλα κράτη-μέλη τα οποία δεν το λένε δημοσίως, αλλά το εκφράζουν ε, εμέσως στην πολωνική κυβέρνηση. Δεν μπορεί λοιπόν να μην το γνωρίσετε, να το ξαναπώ. Ας προσπαθήσουμε να λύσουμε το πρόβλημα, ε, όχι με τιμωρητικό τρόπο, αλλά προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τους Πολωνούς να πάνε ξανά στο σωστό δρόμο του σεβασμού της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Έχετε μια πολιτική εντολή που λάβατε από τους ψηφοφόρους σας. Μπορείτε κι εσείς να το κάνετε. Δεν χρειάζεται να επιτεθείτε στο κράτος δικαίου ε, μην υπαναχωρήσετε ως προς τις βασικές αξίες της Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιτρέψτε μας να κάνουμε αυτό το διάλογο με τους υπουργού σα Εγώ όλη την ημέρα Α, ας μην λέω 24 ώρες το 24ωρο στα αγγλικά, γιατί κάποιος νόμιζε την περασμένη φορά ότι είχα αναφέρει την ημερομηνία 24 ωρο στα αγγλικα γιατι κάποιο Τέλος πάντων εβδομου Τέλο παντων ηθελα να πω ότι νυχθημερών αγωνίζομαι να έχω διάλογο με, τους, ε, ε, ε, με την πολωνική κυβέρνηση, γιατί πρέπει να το λύσουμε αυτό το πρόβλημα ως Ευρώπη. Αν δεν διατηρήσουμε το κράτο δικαίου στην Ευρώπη, Ευρώπη τότε θα χάσουμε τις βασικότερες αξίες Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συνεργασία από αυτόν δεν θα επηρεάσει μόνο την Πολωνία αυτό, αλλά όλα τα κράτη-μέλη, όλους μας. Δεν ζούμε απομονωμένοι, είμαστε πάρα πολύ συνδεδεμένοι μεταξύ μας για να μπορούμε να αφήνουμε τέτοια ζητήματα να εξελίσσονται τόσο άσχημα. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Ολοκληρώνουμε λοιπόν έτσι τη συζήτηση με τον Αντιπρόεδρο. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε και την ομάδα σας. Ευχαριστώ όλους.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 Κοιτάξτε θα περάσουμε στο 5 αλλά περιμένουμε ακόμα την κυρία Μακοβέη. Μπορώ να μιλήσω με κάποιον από τους βοηθούς των συντηρητικών παρακαλώ. Uh, Mrs. Stevens, just seeing if Mrs. Uh, is she here? No, no, no, but she will come. Uh, I'm just so, uh, um, I'm just wondering if Mrs. Stevens uh, would, would. Κυρία Stevens, θα θέλατε να πάρετε το λόγο πρώτα. Θα τελειώσουμε με το σημείο 5 για το επόμενο ε, πολιετές, περιμένοντας την κυρία Μακοβέη. Φαίνεται ότι έχει καθυστερήσει λίγο. Οπότε η κυρία Στίβενς θα παρουσιάσει την πρότασή της, πρόταση γνωμοδότησής της. Χέλγκα, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα αντικαταστήσω μάλλον την κυρία Μάκοβε η οποία έρχεται, αλλά... Συνάδελφοι, σας καλωσορίζω λοιπόν για την παρουσίαση της γνωμοδότησης για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό μετά το 2020. Οι βασικές μου προτάσεις για τους τομείς που θα καλύπτει η ΛΥΜΠΕ είναι οι εξής. Πρώτον, ζητώ τον διαχωρισμό του ασύλου από τα προγράμματα για τα σύνορα και τη δικαιοσύνη σε διαφορετικά κεφάλαια που να ανταποκρίνονται στα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον σεβασμό του κράτους δικαίου, την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη. Τα θέματα αυτά δεν μπορεί να καλύπτονται από τα υπάρχοντα μέσα που είναι περιορισμένα. Θα πρέπει να περιλαμβάνονται και σε μελλοντικά μέσα όπως τα Ταμεία Συνοχής ή και νέα μέσα όπως το Ταμείο για την Ασφάλεια. όλες οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες στον τομέα των εσωτερικών υποθέσεων και της δικαιοσύνης θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα χρήσης των καταπιστευμάτων αυτών. Θεωρώ επίσης ότι τα διαφθρωτικά ταμεία θα πρέπει να συνεχιστούν μετά το 2020 και κάποια από αυτά όπως το κοινωνικό θα πρέπει να αντιμετωπίσουν προγράμματα για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης των, κράτων, των εγκλημάτων μίσους και θα ήθελα επίσης να υπάρξει περαιτέρω χρηματοδότηση για τον τομέα της μετανάστευσης για να αποφύγουμε αυτά τα οποία συνέβησαν κατά τη διάρκεια του ισχύοντος πολιετούς δημοσιονομικού. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε μεγαλύτερη συνοχή ανάμεσα στη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού, του στόχους του προϋπολογισμού και τις μετακινήσεις ανάμεσα στις προτεραιότητες και τις δαπάνες. Πιστεύω ότι η διεύρυνση της χρήσης των καταπιστευμάτων απαιτεί το 100% των ποσών αυτών να περιλαμβάνονται στον κοινοτικό προϋπολογισμό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να είναι σε θέση να ελέγξει τα ποσά αυτά όχι μόνο για την δημιουργία τους αλλά και για την χρησιμοποίησή τους στη συνέχεια. Έκτον, το ισχύον δημοσιονομικό μόνο το 1% καλύπτει δαπάνε Σέγγεν όπως πολιτικές για το άσυλο, μετανάστευση, έλεγχο συνόρων και εσωτερική ασφάλεια. Νομίζω ότι το ποσοστό αυτό θα πρέπει να αλλάξει σύμφωνα με τις προτεραιότητες τις οποίες έχουμε πλέον σήμερα. μου υποστηρίζω πλήρως ε, των ε, εξωτερικών υπηρεσιών για τα θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων και ε, στοχεύουμε στην καλύτερη κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών. Η ανεπαρκής χρηματοδότηση υπηρεσιών όπως το Eurojust, το CIPOL και η Europol είναι κάτι το απαράδεκτο. Η νέα εντολή του Frontex θα απαιτήσει και μετά από το 2020 περαιτέρω μορφές χρηματοδότησης. Να υπενθυμίσω εδώ την ανάγκη που υπάρχει για τους κατάλληλους πόρους έτσι ώστε να καλυφθούν όλα αυτά τα προγράμματα. Υπογραμμίζω την σημαντικό ρόλο του ίδιου Λίσα και ζητώ την γρήγορη εφαρμογή του συστήματος εισόδου-εξόδου όπως επίσης και του συστήματος πληροφόρησης και ενημέρωσης έτσι ώστε ε, να υπάρξει ανταλλαγή ε, ε, τεκμηρίων για ποινικέ υποθέσεις στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επίσης θα πρέπει να υπάρξουν οικονομικές κυρώσεις εις βάρος των κρατών μελών που δεν σέβονται το κράτος δικαίου. Η κατάσταση σήμερα στην Ευρώπη δεν είναι ικανοποιητική οι κυβερνήσεις οι οποίες δεν σέβονται το κράτος δικαίου και την δημοκρατία δεν μπορούν να παραβιάζουν τους κανόνες αυτούς χωρίς να υπάρχουν συνέπειες εις βάρος τους. Σας ευχαριστώ Χέλγα. Η Σιλβή. Εγώ δεν αντικαθιστώ κανέναν. Κατάλαβα, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Μακοβέη. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό θέμα για η χρηματοδότηση των πολιτικών αυτών μετά το 2020 είναι καθοριστική για το μέλλον της Ένωσης και θα πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειες της η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, εγώ σαν σκιώδης Έχω εμείνει στα θέματα της μετανάστευσης. Υπάρχουν κάποια θέματα χαίνοντα και για μετά το 2020 λόγω των κλιματολογικών και δημογραφικών συνθήκων. Δεύτερον, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να καθορίσουμε καλύτερα τις ανάγκες χρηματοδότησης των εξωτερικών υπηρεσιών και τρίτον θα προσπαθήσω να πάρω μέρος στη διευκρίνηση της παραγράφου 7 για την επιβολή οικονομικών κυρώσεων εις βάρος των κρατών μελών που δεν σέβονται ε, το κράτος δικαίου έτσι ώστε να μην πάρουμε αποφάσεις εις βάρος των πολιτών. Λοιπόν, αυτά. Αυτά θα προσπαθήσω να κάνω σαν σκιώδης. Ευχαριστώ Σιλβί. Δεν ξέρω αν κάποιος θέλει το λόγο. Αν όχι, η κυρία Μακοβέη κατάφερε να έρθει. Ε, μπορείτε να κάνετε κάτι, να πείτε κάτι μάλλον, να κάνετε μια παρουσίαση. Ευχαριστώ. Δυστυχώς ε, δεν ήταν δυνατό να με περιμένετε. Ε, ερχόμουν από το αεροδρόμιο και ευτυχώς η Έλγα ήταν αρκετά ευγενής και μίλησε εκ μου. Είναι σημαντικό τα διαφθορτικά ταμεία να συνεχιστούν και μετά το 2020 και κάποια ταμεία όπως το Κοινωνικό Ταμείο να αντιμετωπίσουν την κάλυψη των προγραμμάτων για την ξενοφοβία, την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και εγώ ζητώ περισσότερα χρώματα, χρήματα συγγνώμη, για θέματα που άπτονται του μηχανισμού ευελιξίας του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού όπως και στο ισχύον πολιετές δημοσιονομικό. Θέλουμε μεγαλύτερη συνοχή ανάμεσα στην χρηματοδότηση του προϋπολογισμού και τους στόχους που έχουμε θέσει σε πολιτικό επίπεδο. σεβόμενοι τις ε, αλλαγές των προτεραιοτήτων της Ένωσης. Η διεύρυνση της χρήσης των καταπιστευμάτων σημαίνει ότι το 100% των χρημάτων αυτών θα προέρχονται από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό και ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι σε θέση να εφαρμόσει τον ελεγκτικό του ρόλο. Όχι μόνο σε σχέση με την δημιουργία των ταμείων αυτών, αλλά και σε σχέση με την λειτουργία τους. Τα θέματα αυτά τα είχαμε συζητήσει και στα πλαίσια της συζήτησης για το βρώμικο χρήμα και η άποψή μου η προσωπική είναι ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών είναι η 10η Νοεμβρίου, 12η Μεσημβρινή. Λοιπόν, διακόπτουμε μέχρι τις ψηφοφορίες οι οποίες θα αρχίσουν σε 10 λεπτά. 6 παρατέταρτο.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 να έχετε έτοιμες τις ε, κάρτες ε, ψηφοφορίας σας. Ευχαριστώ. Ξέρω, Δευτέρα απόγευμα είναι, το καταλαβαίνω, αλλά έχουμε πολλές ψηφοφορίες. Παρακαλώ, καθίστε. Ευχαριστώ. Colleagues, everyone ready? I see everyone is not ready, so Παρακαλώ καθίστε. Okay, colleagues, we have... Συνάδελφοι, τέσσερις ψηφοφορίες έχουμε. Πριν περάσουμε στην ψηφοφορία, ευχαριστώ Μόνικα, ευχαριστώ πολύ. Έχετε καθίσει όλοι, όλοι στην τάξη. Ωραία. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ μην κάνετε χειρονομίες εκεί στο βάθος. Λοιπόν, η πρώτη ψηφοφορία είναι κάπως περίπλοκη, οπότε παρακαλώ λίγη ησυχία. Έχετε καθίσει, πρέπει να σας εξηγήσω το πρώτο σημείο που έχουμε να ψηφίσουμε. Μπορεί να είναι και λίγο τσίμα-τσίμα η ψηφοφορία, οπότε παρακαλώ καθίστε. Θέλω όλοι να έχετε καθίσει και να με προσέχετε. Παρακαλώ, τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, παρακαλώ καθίστε και βάλτε την κάρτα σας στη σχισμή. Θα καταλάβετε σε λίγο γιατί. Okay, right. If coordinators are happy that every... Λοιπόν, αν ε, οι συντονιστές ε, είναι ευτυχείς ότι όλοι έχουν προσέλθει, τόσο το καλύτερο. Λοιπόν, είπα κάτι στην αρχή της συνεδρίασης, όμως οι περισσότεροι δεν ήσασταν εδώ, γιατί ήμασταν λίγοι στην αρχή της συνεδρίασης σήμερα. Λοιπόν, είχα πει ότι η έγκριση της απόφασης των συντονιστών θα τις ψηφίσουμε τώρα, πριν από τις ε, ψηφοφορίες τις άλλες. Λοιπόν, ακούστε με, μήπως δεν γνωρίζετε την κατάσταση. Ακούστε με παρακαλώ. Γι' αυτό χτυπάω το σφυρί μου. Συγγνώμη, πονάω ο λαιμός μου και πρέπει να μιλάω χαμηλόφωνα. Ακούστε με λοιπόν. Οι συντονισμένε μα ε, συνεδρίασαν στι 20 Οκτωβρίου και συζήτησαν τι αντιπροσωπείε εντό Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει το άρθρο 205 του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το ζήτησαν ε, οι πράσινοι, ο πράσινο συντονιστή. Πρέπει να ψηφίσουμε λοιπόν την εξή σύσταση για επίσημη έγκριση από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Η σύσταση λοιπόν είναι η εξή. Ε, δυνάμει του άρθρου 205 σύσταση συντονιστή και οι συντονιστές μπορούν να θέσουν αυτό το θέμα σε ψηφοφορία σε ολόκληρη την Επιτροπή. Η σύσταση είναι Λοιπόν, κοιτάξτε με, η σύσταση είναι να μην στείλουμε αποστολή στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας στο πλαίσιο της ειδικής έκθεσης για την κατάσταση στην Ουγγαρία δυνάμει του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου της 17ης Μαΐου 2017. Έλαβα ένα αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία ε, βάσει του κανόνα 308 από τους σοσιαλδημοκράτες, ε, ε, την ΚΟΕ και τους πράσινους, οπότε μπορούμε να κάνουμε ονομαστική ψηφοφορία επ' αυτού. Λοιπόν, θα ψηφίσουμε ως οξύ. Παρακολουθήστε με πολύ προσεκτικά. Αν δεν θέλετε να γίνει αποστολή αντιπροσωπείας της ΛΥΜΠΕ στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, θα πατήσετε το πράσινο κουμπάκι, υπέρ. Αν δεν το καταλάβατε και δεν το κάνετε σωστά, μην με κατηγορήσετε. Αν θέλετε να πάει μια αντιπροσωπεία στην Ουγγαρία, τότε θα πατήσετε το κόκκινο κουμπί που είναι κατά. Αυτό είναι, δεν είναι πολύ διαστητικό γι' αυτό το λέω. Έτσι έχει διατυπωθεί η σύσταση, δεν φταίω εγώ. Εγώ δεν θα έγραφα τίποτε έτσι με αρνητική διατύπωση, αλλά πάση περιπτώσει. Αν δεν θέλετε λοιπόν να πάει η αντιπροσωπεία της Λίμπε στην Ουγγαρία, θα πατήσετε το πράσινο και αν θέλετε να πάει, θα πατήσετε το κόκκινο κατά. Εντάξει, έναρξη ψηφοφορίες λοιπόν, ψηφίστε. Εντάξει, το καταλάβατε όλοι. Το καταλάβατε όλοι. Ωραία, έναρξη ψηφοφορία ηλεκτρονικής. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας λοιπόν. 30 υπέρ, και 21 κατά καμία αποχή. Λοιπόν, άρα να μην πάει αντιπροσωπεία στην Ουγγαρία. Ωραία, εντάξει, ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε τώρα στις ε, ψηφοφορίες και αρχίζουμε με με την έκθεση 2017 για την Ιθαγένεια Ευρωπαϊκή Ένωση ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών σε μια ένωση δημοκρατικής αλλαγής. Τσάμπα Σόγκορ είναι ο συντάκτης γνωμοδότησης. Κύριε Σόγκορ, θέλετε να πάρετε το λόγο πριν την ψηφοφορία. Όχι. Ωραία. Περνάμε λοιπόν. Τροπολογία 60. Έναξη ψηφοφορία. Πέρας. εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10, έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 11, έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 14, έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 23. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Ε, συγγνώμη, τροπολογία 68. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 69. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται. 70. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 13. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 72. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 3. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβασ... Ε, τροπολογία 76 έναρξη ψηφοφορίας. Ζητώ συγγνώμη συνάδελφοι, λέει ο Πρόεδρος. Ξέχασα την συμβιβαστική 17. Ευχαριστώ πολύ κυρία Σίπελ. Συμβιβαστική 17 λοιπόν. Έναρξη ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα, συγκρίνεται. Τροπολογία 76, έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 21. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 19. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 12. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 15. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. 90. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται. 91. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 92. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 93. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρασε. Αγκρίνεται. Συμβιβαστική 22. Έναρξη. Πέρας. Αγκρίνεται. Συμβιβαστική 16. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Αγκρίνεται. Συμβιβαστική 18. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 103. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 106. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. 107. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. 110. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 20. Έναρξη έναρξη Πέρας. Εγκρίνεται. 115. Έναρξη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 117. Έναρξη ψηφοφορία. Πέρασε εγκρίνεται. 118 έναρξη ψηφοφορίας. Πέρασε. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα σε αιτιολογικές σκέψεις και αναφορές, ε, όλες μαζί τροπολογίες 1 έως 3 έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται συμβιβαστική 1 έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται τροπολογίες 6 με 22 όλες μαζί έναρξη ψηφοφορίας. Πέρασε. εγκρίνονται. Συμβιβαστική 2. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρασε. Εγκρίνεται. 24. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. 29. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 5. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. 32. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 34. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται. 36. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. 39. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται. 43. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Κάποιος φώναξε όχι. Τροπολογία 47. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Γκρίνεται. Όλες μαζί 51 ως 59. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Γκρίνονται. Και τώρα ψηφίζουμε το κείμενο όπως έχει τροποποιηθεί με ονομαστική ψηφοφορία. Έναρξη ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται 44 ψήφοι υπέρ, 6 ψήφοι κατά, 3 αποχές. Συγχαρητήρια στον κύριο Σόγκορ. Okay, the draft report now, colleagues, on the proposal for a regulation of the Parliament and Council. Πρόταση κανονισμού, λοιπόν. Εισηγητής, ο Χέρον Λένερ. Θέλετε το λόγο πριν από την ψηφοφορία, κύριε Λένερ. Όχι, περνάμε αμέσως στις ψηφοφορίες, λοιπόν. Τροπολογία 30. Πέρας της ψηφοφορίας απερίφθη. Συμβιβαστική 1. Πέρας. Δεκτή. Συμβιβαστική 2. Πέρας. Δεκτή. 132. Ψηφίζεται. Πέραση της ψηφοφορίας. Δεκτή. Συμβιβαστική 3. Ψηφίζεται. Πέραση της ψηφοφορίας. Δεκτή. Ομαδικά 121, 122, 162 και 50 ψηφίζεται. Πέρας. Δεκτή. Συμβιβαστική 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας τις ψηφοφορίες. Δεκτή προφορική τροπολογία των σοσιαλιστών. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απερίφθε. Συμβιβαστική 5 ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή. 127 ψηφίζεται. Τέλος. Απερίφθη. 20 ψηφίζεται. Πέρας. Δεκτή. 131 ψηφίζεται. Πέρας. Απερίφθη. 135 ψηφίζεται. Πέρας. Απερίφη. 137 και 61 από κοινού ψηφίζεται. Πέρας. Απερίφθη. Συμβιβαστική 6 ψηφίζεται. Πέρας. Δεκτή. Συμβιβαστική 7 ψηφίζεται. Πέρας. Δεκτή. 155 ψηφίζεται. Πέρας. Απερίφη. 156 ψηφίζεται. Πέρας. Δεκτή. Συμβιβαστική 8 ψηφίζεται. πέρας. Δεκτή. 28 ψηφίζεται. Πέρας. Δεκτή. 163 και 83 ψηφίζεται. Πέρας. απερίφθη

167 ψηφίζεται. Πέρας. απερίφη. 29 ψηφίζεται. Πέρας. Δεκτό. 168 ψηφίζεται. Πέραση φοφορία Δεκτή. 32 ψηφίζεται. Πέραση. Απερίφθη. 35 άρχεται. Πέρας. Απερίφθη. 36 άρχεται. Πέρας. Απερίφθη. Συμβιβαστική εννέα, Ψηφίζεται. Πέρας. Δεκτή. 42. Ψηφίζεται. Πέρας. Απερίφθη.

Πέρας. Απερίφθη. 60 άρχεται. Πέρας. Δεκτή. 62 άρχεται. Πέρας. Απερίφθη. 68 άρχεται. Πέρας. Απερίφθη. 69 άρχεται. Πέρας. Δεκτή. 77 ψηφίζεται. Πέρας. Απερίφθη. 78 και 80 ταυτόσημες ψηφίζεται. Πέρας. Απερίφθη. Άφετε 7 ψηφίζεται. Τέλος. Απερίφθη. 81 ψηφίζεται. Τέλος. Απερίφθη. 82 ψηφίζεται. Τέλος. Απερίφθη. 87 ψηφίζεται. Πέρας, απερίφθη. Εννέα ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή. Άφετ οκτώ ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή. Τροποποιημένο κείμενο. Ονομαστική κλίση ψηφίζεται. Πέρας της ψηφοφορίας 44 υπέρ 5 κατά. Ψηφοφορία για την έναρξη διαπραγματεύσεων. Ψηφίζεται. Πέρας. 42 υπέρ 5 κατά 4 αποχές. Συγχαρητήρια στον κύριο Λένερς. Καλώς συνάδελφοι. Προχωρούμε στο σχέδιο έκθεση Συμβουλίου και Κοινοβουλίου για την χρήση του συστήματος πληροφοριών Σέγγεν στον τομέα των συνοριακών ελέγχων για ε, κατάργηση της, ε, του κανονισμού 515 και της οδηγίας 1987-2006. Ε, ο Κάρλος Κουέλιο είναι ο εισηγητής. Θέλετε το λόγο, παρακαλώ. Ναι, Πρόεδρε, σύντομα για να ευχαριστήσω όλους. Ξέρω ότι ήταν πραγματικά πολλή δουλειά που πρέπει να κάνουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά έχουμε τους συμβούλους μας, τους βοηθούς, τη γραμματεία που βοήθησαν. Η δουλειά έγινε πολύ ευχάριστα, σε πολύ καλό περιβάλλον. Και θέλω απλώς να πω ότι όλοι μας ή τέλο πάντων οι περισσότεροι από εμά θέλουμε να προστατεύσουμε τη Σέγγεν και την ελευθερία ε, κυκλοφορίας, αλλά θέλουμε να το κάνουμε αυτό με ασφάλεια. Και με αυτό το νομοθετικό κείμενο αυτό προσπαθούμε να επιτύχουμε. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Κουέλιο. Πάμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. Τροπολογία 22 και 23 μαζί. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το άρθρο 3, Αρχητη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε από κοινού 32 έως 36. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνονται. Ψηφίζουμε συνολικά την 37 και την 38. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 223. 224, ε, συγγνώμη. Ε, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 225. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το άρθρο 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 228. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 236. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 42. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το άρθρο 10. αρχήτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 46. αρχή ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ε, συμβαστική για, την, για το άρθρο 12. αρχή ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 245. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 2.47. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το άρθρο 14. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε από κοινού την 50 έως 56. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνονται. Συμβαστική για το άρθρο 16. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 61. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το άρθρο 18. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 259. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Αχ, ψήφισα λάθος, αλλά εντάξει δεν αλλάζει το αποτέλεσμα. Συγγνώμη στο συντονιστή μου. Ξέρετε, προσπαθώ να διεξάγω και τις ε, ε, ψηφοφορίες και να ψηφίσω ταυτόχρονα. Λοιπόν, ε, συμβαστική για το άρθρο 19. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το άρθρο 20. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το άρθρο 21. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική για το άρθρο 22. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το άρθρο 23. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το άρθρο 23α. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το άρθρο 24. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το άρθρο 26. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το άρθρο 27. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το 27α. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το άρθρο 28. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το άρθρο 29. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το άρθρο 30. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το άρθρο 31. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το άρθρο 32. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ε, άρθρο 34. Συμβαστική για το άρθρο 34. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το άρθρο 35. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το άρθρο 36. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 383. Πέρας. Απορρίπτεται. Ε, τροπολογία 34. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική για το άρθρο 38. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το άρθρο 39. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το άρθρο 40. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το άρθρο 41. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το άρθρο 42. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 405. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 406. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική για το άρθρο 46. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το άρθρο 47. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το άρθρο 48. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το άρθρο 49. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το άρθρο 50. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το άρθρο 51. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το άρθρο 52. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το άρθρο 53. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το άρθρο 54. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το άρθρο 54α. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το άρθρο 58. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Ε, αιτιολογικές σκέψεις. Ε, συμβαστική για, το αιτιολογική, για την αιτιολογική σκέψη 6. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική για την αιτιολογική σκέψη 6α. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική για την αιτιολογική σκέψη 7. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική για την αιτιολογική σκέψη 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική για την αιτιολογική σκέψη 9 και 9α. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική για την αιτιολογική σκέψη 11. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συμβαστική για την ιδεολογική σκέψη 12. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική για την ιδεολογική σκέψη 13. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική για την ιδεολογική σκέψη 15. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση για την αιτιολογική σκέψη 16. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική για την αιτιολογική σκέψη 17. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 160. Πέρας πληροφορία. Εγκρίνεται. Συμβαστική για την αιτιολογική σκέψη 18. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική για την ετουλική σκέψη 20. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική για την ετουλική σκέψη 21. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική για την ετουλική σκέψη 23. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική για την ειδηλική σκέψη 24. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική για την ειδηλική σκέψη 25. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική για την ειδηλική σκέψη 26. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική για την αιτιολογική σκέψη 27. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική πρόταση για τις ε, σκέψει σκέψεις 28, 28α, 28β, 28γ και 28δ. Πέρας εγκρίνονται. Συμβαστική για, το, για την Ανατολική Σκέψη 31. 31. Πέρας της Εγρίνεται. εγκρίνεται. Συμβαστική για την αιτιολικη σκεψη σκέψη 32α. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το ενετολική σκέψη 33. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική για την ενετολική σκέψη 34. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική για την αιτιολογική σκέψη 35. Άρχεται η ψηφοφορία. Μπορούν οι συντονιστές να μην φωνάζουν τόσο δυνατά τι πρέπει να ψηφίσουν οι υπόλοιποι. Πέρας ψηφοφορίας και εγκρίνεται η 35. Συμβαστική για την αιτιολογική σκέψη 36. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 194 τροπολογία. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική για την αιτιολογική σκέψη 37. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 200. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική για την ετολική σκέψη 38. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική για την ετολική σκεψη σκέψη 38α. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική για την ετολική σκέψη 40. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική για την αιτιολογική σκέψη 40α. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική για την αιτιολογική σκέψη 42. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Άφετ 6. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 205. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το είναι τελική σκέψη 53. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Αφετεπτά, 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το κείμενο όπως ε, τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 45 ψήφοι υπέρ, 3 ψήφοι κατά και 5 αποχές. Και η ψηφοφορία για την απόφαση να μπούμε σε διαπραγματεύσεις. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 43 ψήφοι υπέρ, 5 ψήφοι κατά, 4 αποχές. Συγχαρητήρια κύριε Κοέλιο. Last vote, colleagues, last one. Τελευταία ψηφοφορία, συνάδελφοι, τελευταία. Be patient. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και την υπομονή σας. Είμαστε στην τελευταία ψηφοφορία. Colleagues, we'll have to go quite fast, interpreter. Οι διερμηνείς πρέπει να αποχωρήσουν, οπότε πρέπει να πάμε πολύ γρήγορα. Πολύ γρήγορα. Αν θέλετε σιγά σιγά. Εντάξει, γρήγορα τότε θα πάω. Κύριε Κοέλιο, θέλετε να πάρετε το λόγο. Σας χειροκρότησαν όμως αρκετά. Λοιπόν, σας πειράζει να ψηφίσουμε απευθείας τροπολογία 30. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρασε. Α, τι ψηφίζουμε, ναι, συγγνώμη, ξέχασα να το πω. Αυτό πάω από τον τίτλο. Πέρας ψηφοφορίας πάντως. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική άρθρο 3 ορισμοί. Έναρξη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 41. Άρχεται η ψηφοφορία. Μα μισό λεπτό. Συνάδελφοι, συγγνώμη. Κουράστηκα και εγώ, ναι, μη βαράτε. 41 μέχρι 45 από κοινού. Έναρξη ψηφοφορία. Πέρασε. 46 και 47 μαζί. Έναρξη ψηφοφορία. Πέρασε. Αγκρίνεται. 267. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 268. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική άρθρο 8. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. 271. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρασα. Εγκρίνεται. 280 έναρξη. Πέρασα. Εγκρίνεται. 51 έναρξη ψηφοφορίας. Πέρασα. Εγκρίνεται. Συμβεβαστική άρθρο 10. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρασα. Εγκρίνεται. Τροπολογία 55. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική άρθρο 12. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 289. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρασε. Εγκρίνεται. 292 έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός άρθρο 14. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. 60 έως 65 όλες μαζί. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνονται. Συμβιβαστική άρθρο 16. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 70. Έναρξη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική άρθρο 18. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 305. Έναρξη. 305. Πέρασε. Πορύπτεται. Συμβαστική άρθρο 19. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρασε. Εγκρίνεται. Όλες μαζί από 315 μέχρι 198. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. Όλες μαζί και πάλι από 316 μέχρι την 199 έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική άρθρο 20. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρασε. Γκρίνεται. Συμβαστική άρθρο 21. Έναρξη. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συμβαστική άρθρο 22. Έναρξη. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική άρθρο 23. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική άρθρο 23A. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική άρθρο 24. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική άρθρο 26. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική άρθρο 32. Έναρξη. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική άρθρο 33. Έναρξη. Πέρασε. Εγκρίνεται. Ε, συμβιβαστική άρθρο 36. Έναρξη. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 391. Έναρξη. Πέρασε. Απορρίπτεται. 396 έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική άρθρο 37. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική άρθρο 38. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική άρθρο 39. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική άρθρο 40. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. 418. Πρώτο τμήμα. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική άρθρο 40, δεύτερο τμήμα. Έναρξη. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συμβαστική άρθρο 41, έναρξη. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συμβαστική άρθρο 42, έναρξη. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική άρθρο 43. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική άρθρο 44. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική άρθρο 45. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική άρθρο 46. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική άρθρο 47. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική άρθρο 48. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική άρθρο 49. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική άρθρο 51. Έναρξη. 51. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική άρθρο 52. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική άρθρο 53. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική Α, συγγνώμη. 5.26. Έναρξη. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συμβαστική άρθρο... That doesn't fall. There is none. Να we do vote 526. ψηφίζουμε την 526. Πρέπει να την ψηφίσουμε την 526. Και την ψηφίσαμε μόλις. Εντάξει. Ωραία. Τέλεια. Καλώς. Μήπως μπορούμε να ελέγξουμε την ε, ψηφοφορία γιατί εδώ λέει ότι εκπίπτει με τον ε, συμβιβασμό. Ναι, πραγματικά προκαλεί σύγχυση ο κατάλογος ψηφοφορία, αλλά μήπω θέλετε να ξαναψηφίσουμε επειδή υπάρχει αυτή η σύγχυση. Εντάξει. Λοιπόν, να ξαναψηφίσουμε. Θα ψηφίσουμε την 526 ξανά. Ψηφίζουμε λοιπόν την 526. Παρακαλώ ψηφίστε. Επαναλαμβάνουμε την ψηφοφορία γιατί εδώ ε, είναι κάπως λάθος η ένδειξη στον κατάλογο ψηφοφορίας και δημιουργήθηκε σύγχυση. Λοιπόν, απορρίπτεται. Συμβιβαστική άρθρο 55. Έναρξη ψηφοφορίας. 55. Ψηφίζουμε το άρθρο 55. Συν και πάλι. Πέρας. Γκρινέτ. Συμβαστική άρθρο 56. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική άρθρο 57. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική άρθρο 58. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. συμβαστική άρθρο 59. Έναρξη. Μισό λεπτό. Μετά το 58 δεν έκλεισε η ψηφοφορία. Πάμε πολύ γρήγορα. Μας προδίδουν οι μηχανές. Colleagues, could you just... Colleagues... Συνάδελφοι, λίγη υπομονή δείξτε παρακαλώ. Okay. Okay, colleagues, please just be... Συνάδελφοι, λίγη υπομονή παρακαλώ. I'd like to thank colleagues. Συνάδελφοι, συγγνώμη, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διερμηνείς που θα παραμείνουν μέχρι το τέλος της ψηφοφορίας, ακόμη 10 λεπτά. Τους ευχαριστώ λοιπόν. Πού ήμασταν, στο άρθρο 59. Το ψηφίσαμε το 59. να ψηφίσουμε το 59. Για όσους φεύγουν, σχεδόν έχουμε τελειώσει. Άρθρο 59 λοιπόν, συμβαστική έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 550 έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται. 551 έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική άρθρο 63 έναρξη. Πέρας. Τι έγινε. Τι έγινε με την 63. Yeah, but, but it's not. The vote is closed. What's happening? Έχει ολοκληρωθεί η ψηφοφορία. Τι έγινε, κάτι συμβαίνει εδώ με το, με τη μηχανή, με το μηχάνημα. Λοιπόν, ψηφίζουμε και πάλι την 63. Κάτι γίνεται εδώ. Δεν δουλεύει καλά το μηχάνημα. Λίγη ησυχία παρακαλώ, συνάδελφοι. Άρθρο 63 και πάλι. Άρθρο 63 ψηφίζουμε.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 όλες τις υπόλοιπε συμβιβαστικέ μπορούμε να τι ψηφίσουμε όλες μαζί. Ρωτάω τον εισηγητή. Ε, κοιτάω τον εισηγητή. Να μα πει. Λοιπόν. Λοιπόν. Πατήστε λοιπόν το πράσινο κουμπάκι για όλες μαζί τις συμβιβαστικέ τροπολογίες. Έναρξη ψηφοφορία Εκτός αν δεν θέλετε Oh, I knew that was going to happen. Ξέρα ότι θα γίνει αυτό. Εντάξει, εντάξει, εντάξει, υπομονή. Να συνεχίσουμε λοιπόν. Λοιπόν, στην 64 είμαστε λοιπόν. Συμβιβαστική για το 64, έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Γκρίνεται. 65. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Άρθρο 66. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Άρθρο 68, λέει ο πρόεδρος. Α, ξέχασα την 67. Δεν το συγγνώμη. Άρθρο 67, έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Άρθρο 68. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Γκρίνεται. Άρθρο 69. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Γκρίνεται. 70. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Άρθρο Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρασε. Εγκρίνεται. Άρθρο 71. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Άρθρο 71A. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Άρθρο 75. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Πάμε στι αιτιολογικές αναφορέ. Λοιπόν, για το 6, έναρξη ψηφοφορία. πέρας. Εγκρίνεται. Για το 6, εναρξη ψηφοφορία. ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. 6A, έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. 7, έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Οκτώ. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Εννέα και εννέα ει. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Έντεκα. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας εγκρίνεται 12. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται 13. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται 15. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται 16. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται 17. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. 18. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. 191. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική για την αιτιολογική σκέψη 19. Συγγνώμη, τι θέλετε για την 191. Ποιο είναι το πρόβλημα. Τι έγινε. you, do I have permission to take the vote again? Μπορούμε να ξαναψηφίσουμε παρακαλώ. Κοιτάξτε, αν πρέπει να ξανακάνουμε την ψηφοφορία, πρέπει να μου το επιτρέψει όλη η Επιτροπή. Αν είναι λάθος, είναι διαφορετικό, Τζούντιτ. Αν είναι ένα αίτημα για επανάληψη ψηφοφορίας, είναι αλλιώς. Yeah. In was the machine not working in the middle of the Okay, that's fine. Is working now? Δεν δούλευε δηλαδή το μηχάνημα κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Μήπως μπορείτε να πάτε κάπου αλλού να καθίσετε τότε, γιατί πάλι θα έχετε αυτό το πρόβλημα. Νομίζω ότι ο κόσμος απλώς θέλει να φύγει. Όλοι θέλουμε να φύγουμε. Άννα, μήπως θες να πασαλούμε την κάρτα σου για να ψηφίσεις και θα δούμε. Λοιπόν, συνάδελφοι, παρακαλώ, υπομονή, υπομονή. Τελειώνουμε, τελειώνουμε. Μερικές σελίδε ακόμη. 191 έναρξη ψηφοφορία. Oh, Oh, well Δουλεύει, μπράβο, μπράβο. Πέρασε. Απορρίπτεται. Well, in a nicer sort of balanced way. Τέλος πάντων, με πιο εξισορροπημένο τρόπο όμως. Λοιπόν, συμβιβαστική για τη βιολογική σκέψη 20, έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική την αιτιολογική 23. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Παρακαλώ, υπομονή και ησυχία. 23. A. Ε, έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. 23A. Ε, έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται 24. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 216. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Αιτιολογική 26. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. 29. Έναρξη. Πέρας. Γκρίνεται. 30. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. 225. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. 32. λογική 32. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. 33. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική για το 34. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Γκρίνεται. Συμβαστική 35. Έναρξη ψηφοφορία. Πέρας. Γκρίνεται. Για το 36 τώρα, συμβαστική έναρξη ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Για το 36A, έναρξη ψηφοφορίας. Πέρασε. Εγκρίνεται. 36B, Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Γκρίνεται. 36C. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. 231. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρασε. Απορρίπτεται. 232 έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. 38 έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. 41. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. 42A. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. 43. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. 44. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. 45. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. 46. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. 47. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται 48. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται 48A. Ε, έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται 50. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται 50A. Ε, έναρξη. Πέρας. Γκρίνεται. 52. Έναρξη. Πέρας. γκρίνεται, 252. Έναρξη. Πέρας. Γκρίνεται. 64. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα το τροποποιημένο κείμενο με ονομαστική κλίση. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. 41 υπέρ, 3 κατά, 4 αποχές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ψηφίσουμε τώρα την απόφαση για την έναρξη διαπραγματεύσεων. Έναρξη. Πέραση. Πέρας, συγγνώμη. Εγκρίνεται 40 ψήφοι υπέρ, 5 κατά, 2 αποχές. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια κύριε Κοέλιο. Τέλος ψηφοφορίας.